Λοιπόν, προσπάθησα να καλέσω όλους αυτούς οι οποίοι ήταν έξω, αλλά δεν τα κατάφερα. Ναι. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία του Γενικού Διευθυντή του κ. Πόλγερ που είναι μαζί μας. Ορισμένοι μπορεί να ρωτήσουν γιατί δεν έχει έρθει η κυρία Ρέντινγκ, μα δεν του καταλαβαίνω. Η κυρία Ρέντινγκ ήταν εδώ το Δεκέμβριο. Και τώρα χρειαζόμαστε αυτόν, ο οποίος σαν υπεύθυνο με την υπό την αιγύδα της κυρίας Ρέντινγκ εκτελεί <clears throat> τις απαραίτητες ενέργειες. Γι' αυτό χαιρετίζω τον κύριο Πόλγκερ και ο κύριος ε, Τάκουλα θέλει να πει κάτι εξ ονόματος του κυρίου Λόκεγκατ αλλά έχετε το maximum τρία λεφτά. Πρέπει να τα πείτε όλα σε τρία λεφτά. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Στάκουλα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε κάθε περίπτωση. Χαίρομαι για την παρουσία του κύριου Πάουλγκερ και θα μας δώσει την άποψή του ο κύριος Λόκεγκάρντ. Και άλλοι συνάδελφοι τον έχουν ήδη γνωρίσει. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά καλά στοιχεία σε αυτή την έκθεση, αλλά δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο σε αυτή την έκθεση. Εμείς είχαμε ζητήσει να παρουσιαστεί μια συνολική στρατηγική και αυτό δεν νομίζω ότι είναι η θέση μονάχα των φιλελευθέρων και η θέση του ΕΛΚ και των ε, σοσιαλιστών και γι' αυτό έχουμε καταθέσει μια σειρά τροπολογιών στην Επιτροπή, στην Επιτροπή Συνταγματικών ε, Υποθέσεων. Δεν θέλουμε λοιπόν να παραμείνει αποσπασματική αυτή η στρατηγική από την πλευρά της Κομισιόν. Αντίθετα θέλαμε μια συνολική στρατηγική θα ήταν χρήσιμο η Επιτροπή μας μαζί με τη Συνταγματική Επιτροπή επομένως καταφέρει να έχει μια κοινή θέση μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σε σύνδεση με το σημείο αυτό ελπίζω ότι μπορεί ο κύριος Πάλουγκερ να μας εκπλήξει και να μας παρουσιάσει μια συνολική και πλήρη στρατηγική αυτό το οποίο λοιπόν έχουν ε, επικρίνει ο κύριος ε, Λόκεργαρτ και άλλοι, τότε δεν θα ισχύει. Ελπίζω παρόλα αυτά ότι η, η παρέμβασή σας θα αντιστοιχεί σε αυτά τα οποία έχει ζητήσει από εσάς η Επιτροπή μας. Ευχαριστώ Χάνου. Για να ελέγξεις ότι πράγματι έτσι θα είναι θα πρέπει να μείνεις εδώ και να παρακολουθείς τις συνεδρίες. Χωρίς μικρόφωνο κύριο Στάκουλα not correct. You cannot report... Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν μπορείς να πεις στο φίλο στο Λόκεργα τι γίνεται άμα φύγεις. Κάποιος θα πρέπει να μείνει στη θέση σου, αλλιώς αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό. Σου έδωσε το λόγο και άμα φύγεις είναι κακό αυτό. Εγώ προσπαθώ να είμαι δίκαια εναντί όλων. Αν θες να διαμαρτυρηθείς για κάτι, θα πρέπει να Γνωρίζει περί πρόκειται. Αυτό ήταν το παρελθόν μου ως δασκάλα. Λοιπόν, μπορείτε να το ξεχάσετε. Κύριε Πάουλγερ, σας δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο. Θεωρώ ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Κοινοβούλιο έχουμε ένα κοινό όραμα να διαβιβάζουμε το μήνυμα της Ευρώπης αποτελεσματικά στους πολίτες της. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι εδώ στην Επιτροπή σας, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερος ε, στο ρόλο μου για πρώτη φορά ως Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας. Σήμερα έχουμε την έκθεση 2012 για την επικοινωνία της Ευρώπης ε, στους πολίτες και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι στην ε, σταθερή βάση συνεργασίας μας ε, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη σχέση, τη σύμπραξη της ε, επικοινωνίας στην Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να εμπιστεύονται τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι στο 15% στοιχείο της Eurostat που είναι πολύ χαμηλό και θα πρέπει να αποδείξουμε στους πολίτες ε, την ε, προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαντώντας συγκεκριμένα ερωτήματα όπως ε, το γιατί χρειαζόμαστε μια οικονομική διακυβέρνηση, τι δικαιώματα έχω εγώ ως Ευρωπαίος πολίτης, τι υποχρεώσεις έχω στην καθημερινότητά μου. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι η Ευρώπη μας είναι η Ευρώπη των πολιτών και για να συνεισφέρουν αποτελεσματικά οι Ευρωπαίοι πολίτες στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να κάνουμε προσπάθειες το 2012 ώστε να αναπτύξουμε τη νέα φάση των επόμενων 24 μηνών. Μόνο αν θέσουμε γερά θεμέλια τώρα μπορούμε να έχουμε επιτυχία στην προσπάθειά μας να γνωστοποιήσουμε τη σημασία της Ευρώπης για τους Ευρωπαίους πολίτες ε, για την ε, δύσκολη περίοδο που μας περιμένει. Υπάρχουν ε, μέσα, αντιπροσωπείες, ε, ιστοσελίδες ε, της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας και όλα αυτά θα αποτελέσουν το επίκεντρο των προσπαθειών μας και θα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να ε, προσεγγίσουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντα μας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το ίδιο ε, είναι αυτό το οποίο ενσωματώνει αυτή τη δέσμευση διότι έχει την δημοκρατική νομιμότητα από τους Ευρωπαίους πολίτες. Ε, αυτή η νομιμότητα προκύπτει από τις ελεύθερες ευρωεκλογές όχι μόνο ε, λοιπόν νομιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά προάγει και κάποια από τα βασικά ιδανικά. Ε, το ποιο είναι υπέλογο σε ποιον, την ελευθερία του λόγου και πολλά άλλα. Ένα λοιπόν βασικό στόχο ε, για το Ευρωπαϊκό Έτο Πολιτών το 2013 θα είναι να κινητοποιηθεί το Ευρωπαϊκό Εκλογικό Σώμα ώστε να συμμετάσχει στι εκλογέ του 2014. Εμείς λοιπόν στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας θα θέσουμε την εμπειρογνωμοσύνη και τα εργαλεία μας στη διάθεσή σας ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση ε, προς το κοινό για τις ευρωεκλογές. Ε, με βάση τα στοιχεία του Ευρωβαρομέτρου θα ασχοληθούμε με το θέμα της ευρωπαϊκής υπηκότητας αλλά αυτό σημαίνει ότι και εσεί, ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να ε, οικειοποιηθείτε αυτή τη διαδικασία και να συνεργάζεστε μαζί μας σε όλα τα στάδια, κατά την προετοιμασία, κατά την εφαρμογή, αλλά και στη συνέχεια. Να σας πω λίγα πράγματα για την διοργανική συνεργασία. Η ομάδα ενημέρωσης ε, σε διοργανικό επίπεδο, η IGI, αποτελεί βασικό πλαίσιο για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε αποτελεσματικά ώστε να διαβιβάσουμε τις προτεραιότητες του IGI, να δημιουργήσουμε την ευρωπαϊκή υπηκότητα, να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ε, συζήτησα το θέμα των ευρωεκλογών με τους δύο νέου αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα επικοινωνία, την κυρία Άννη Ποδηματά και τον κύριο Ότμαν Κάρας. Οι συνεδριάσεις αυτές αποτελούν το πρώτο βήμα σε αυτή την κοινή προσέγγιση. Η IGI, όπως συμφωνήσαμε, θα αποτελέσει βασικό φόρουμ για τη συνεργασία μας και την προετοιμασία των ευρωεκλογών. Τον Ιούνιο του 2011 η διοργανική αυτή ομάδα ζήτησε από όλα τα θεσμικά όργανα να γίνει ένα επιτυχές ευρωπαϊκό έτος πολιτών. Θα υπάρξει μια νέα συνεδρίαση σε διοργανικό επίπεδο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, η οποία θα μας επιτρέψει, και ε, αναφέρομαι σε ολομέλεια της IGI, να καθορίσουμε ε, ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Να περάσω τώρα στην έκθεση που σας παρουσιάζεται σήμερα από την Αντιπρόεδρο Ρέντινγκ. Να διευκρινίσω το εξής επιπλέον. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούμε τι έχει να μας πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε λάβει υπόψη πάμπολε συστάσει από τι εκθέσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα ενημέρωση. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώ θα αναπτύξουμε περαιτέρω τα υφιστάμενα μέσα επικοινωνία που διαθέτουμε, ώστε να έχουμε μεγαλύτερη επικοινωνία σε επίπεδο κρατών μελών, να είναι δηλαδή πιο αποκεντρωμένη η επικοινωνία, ώστε να βελτιωθούν οι πληροφορίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για του πολίτε και του δημοσιογράφου και για να ε, προωθήσουμε έναν πανευρωπαϊκό διάλογο μέσω τη υποστήριξη των μέσων ενημέρωση. Το να υπάρχει λοιπόν καλύτερη επικοινωνία σε επίπεδο κρατών μελών σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους πολίτες, συγκεντρώνοντας ε, την επικοινωνία τοπικοί φορείς ε, γνωρίζοντας την πολιτική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής ε, μας επιτρέπουν να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες των πολιτών. Ιδίω σε πλαίσια οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε να βρούμε τον πιο αποδοτικό ως προς το κόστος τρόπο για να προσεγγίσουμε τους πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι θα εφαρμόσουμε τα μέσα επικοινωνία μας ε, ε, ε, στα κράτη-μέλη συμπράξεις διαχείρισης οι οποίες γίνονται σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί παραδείγματι. Τώρα, στους ευρωπαϊκούς δημοσίους χώρους, τα EPS, εμείς ε, έχουμε αναπτύξει μια ιδανική πλατφόρμα για να συνεργαζόμαστε για κοινέ δραστηριότητες. Υπάρχουν δύο νέα EPS τα οποία προσθέθηκαν το 2011 και έχουμε σύνολο 16 τα οποία έχουν υποδεχθεί ε, περίπου 3 εκατομμύρια Ευρωπαίους πελέτους αποτελούν ε, μοναδική πλατφόρμα για να ε, διεγείρουμε το ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά ζητήματα, ιδιαίτερα σε συστοχευμένες ομάδες όπως για παράδειγμα την νεολαία. Το 2012 θα σημαίνει ότι θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο και θα σταλεί και μια αξιολόγηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ε, δραστηριότητες του 2011 και το φετινό πρόγραμμα εργασία, κατόπιν αιτήματο ε, της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων στην οποία απαντήσαμε. Επίσης υπάρχουν 18 συμπράξει συνεργασία διαχείρισης στα κράτη-μέλη που βασίζονται σε διμερή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κρατών Μελών και αυτά αποδεικνύονται πολύ καλά μέσα για τη συνεργασία. Είναι πολύ καλά επιτόπου, συμμετέχουν οι εθνικές και περιφερειακές αρχές και υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες επικοινωνίες οι οποίες λαμβάνουν περισσότερη πολιτική νομιμότητα και έχουν και παρουσία σε ε, τομεί στου οποίου η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περιορισμένε αρμοδιότητε, όπω για παράδειγμα τα θέματα τη παιδεία. Υπάρχουν επίσης και κάποια εκδηλώσεις οι οποίες προβάλλονται περισσότερο προς τους πολίτες. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι βάσει αυτών όλων των δραστηριοτήτων θα υπάρχει ε, σημαντική αύξηση για όλα τα προγράμματα τα οποία ξεκίνησαν το 2011. Φέτος, οι δραστηριότητες επικοινωνίες που έχουν οργανωθεί θα περιλαμβάνουν και τηλεοπτικά προγράμματα, συζητήσεις ε, και εκπαίδευση ε, διδασκόντων σε ευρωπαϊκά ζητήματα. Να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκή Ένωση για τους πολίτες και τους δημοσιογράφους. Αυτό γίνεται σε καθημερινή βάση. Υπάρχουν τρία βασικά παραδείγματα που καταδεικνύουν ότι υπάρχουν συγκεκριμένε δραστηριότητε. Καταρχά τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Άμεσων Πληροφοριών, τα λεγόμενα ethics. Κατόπιν Υπάρχουν ε, οι γωνιές για τα παιδιά και τους δασκάλους. Αυτές είναι συγκεκριμένες ιστοσελίδες ε, τύπου μέσων δικτύωσης, ε, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Και επίσης υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες για τους δημοσιογράφους. Υπάρχουν περίπου 200 ethics σε όλα τα κράτη-μέλη, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν να προσεγγίσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στους πολίτες της, παρέχοντας ένα άμεσο σημείο επαφής που επιτρέπει στους πολίτες πολίτες να ανακαλύψουν για παράδειγμα ποια είναι τα δικαιώματά τους βάσει της ευρωπαϊκής ε, νομοθεσίας των συνθήκων και του δευτερογενούς δικαίου. επίσης υπάρχει μια προσέγγιση μια στιρίδας στην οποία μπορούν να λάβουν πληροφορίες οι Ευρωπαίοι πολίτες μέσω τηλεφώνου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Άμεσης Επαφής, υπάρχει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών, αλλά και στο διαδίκτυο. Υπάρχει συγκεκριμένη δικτυακή πύλη το τέλος του έτους ε, εκπνέει η προθεσμία των έτηξ που έχουμε και θα πρέπει να αποφασιστεί η χρηματοδότηση για την επόμενη γενεά από το 2013 μέχρι το 2017. Αυτό θα μας διασφαλίσει ότι οι πολίτες θα δουν το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πολλά χρόνια ακόμα. Και τα έτηξ είναι ο τρόπος με τον οποίο εσείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκφράσατε το ενδιαφέρον σας. Έχει συμπεριληφθεί μια τροπολογία στον προϋπολογισμό του 2012 που ζητούσε να συμπληρώσουν τα έτηξ ε, το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, απαντούν στις ερωτήσεις των πολιτών ε, για τις ευρωεκλογές επί παραδείγματι και γι' αυτό ακριβώς αποτελούν βασικό τμήμα της προσέγγισης μας για να διαβιβάζουμε το μήνυμα της Ευρώπης πιο αποτελεσματικά στους πολίτες μας. Επίσης ε, προσεγγίζουμε τους πιο νέους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρσι, ως τμήμα της ατζέντα για τα δικαιώματα των παιδιών, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα Kids Corner που σας ανέφερα. Είναι μια ενιαία θηρίδα όπου υπάρχουν παιχνίδια, ερωτηματολόγια και εύκολες πληροφορίες για τους νέους ανθρώπους. Υπάρχει επίσης μια γωνιά δασκάλων όπου υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό για τις τάξεις των ε, ε, δασκάλων. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να προάγουμε αυτά τα πολύ πολύτιμα μέσα φέτος για να προάγουμε τη συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Επιπλέον εξετάζουμε πέραν ε, των ε, ε, κέντρων τύπου των Βρυξελών για να βρούμε και επαφές στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν σεμινάρια για δημοσιογράφους, για τα νέα μέσα ενημέρωσης. Χρησιμοποιούνται ευρύτατα. Για παράδειγμα, είχαμε δύο επισκέψεις στην Ελλάδα από δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη που επιβεβαιώνουν πόσο χρήσιμα είναι αυτά τα εργαλεία. Επιπλέον μπορούμε να διοργανώνουμε πλέον σεμινάρια οπουδήποτε στον κόσμο για δημοσιογράφους, αλλά το παρόν πλαίσιο επιτρέπει και στα άλλα θεσμικά όργανα, όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να φιλοξενεί αυτά τα σεμινάρια. Υπάρχουν και τα ευρωπαϊκά κέντρα πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, ώστε να γνωστοποιηθούν περισσότερο τα ευρωπαϊκά ζητήματα σε εθνικό επίπεδο. Ε, υπάρχουν αντιπροσωπείες και τα κέντρα ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα οποία θα διοργανώσουν συνεντεύξει τύπου και θα απαντούν από κοινού στις ερωτήσει των δημοσιογράφων. Να περάσω τώρα στην ε, πανευρωπαϊκή συζήτηση μέσω υποστήριξης ε, δικτύων μέσων ενημέρωσης. Μέσω αυτών των ολοκληρωμένων δικτύων ενημέρωσης θα προάγουμε μια συγκεκριμένη συζήτηση για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τους πολίτες με πληροφορίες υψηλής ποιότητας σε ευρύ φάσμα μέσων ενημέρωσης, μέσω της τηλεόρασης, ε, της έντυπης δημοσιογραφίας ε, και του διαδικτύου. Υποστηρίζουμε το Euronews, θα υποστηρίζουμε επίσης και το διαδικτυακό εργαλείο Press Europe και θέλουμε να φέρουμε την ευρωπαϊκή συζήτηση και στις νεότερες γενναίες ε, διασφαλίζοντας ότι θα έχουμε παρουσία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα ληφθούν κανάλιλα μέσα ώστε να συμμετέχουμε εκεί. Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες έρευνες οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι συστηματικά η τηλεόραση είναι το βασικό μέσο ενημέρωσης για τους Ευρωπαίους πολίτες και από εκεί λαμβάνουν τις πληροφορίες τους για την Ευρώπη. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι η τηλεόραση είναι ένα αντικατάστατο μέσο ενημέρωσης και θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες ώστε να προωθήσουμε μια πραγματική συζήτηση για τα ευρωπαϊκά ζητήματα μέσω του Euronews. Το Euronews είναι το βασικό δίκτυο το οποίο ε, μεταδίδει το πρόγραμμά του τώρα σε 20 γλώσσες και δίνει καθημερινά ενημέρωση ε, όπως αποδείχθηκε το 2011. Η συμφωνία πλαίσιο που έχουμε με το Euronews είναι ανοιχτή όχι μόνο για, το Ευρωπαϊκό, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, περιλαμβάνοντας φυσικά και το Κοινοβούλιο. Το 2012, μετά από προτάσεις ε, της έκθεσης που σας ανέφερα για τη δημοσιογραφία και τα νέα μέσα ενημέρωσης, ε, θα περάσει το θέμα της συζήτησης για την Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη, μέσω επεκτάσεων ε, και γλωσσικών αλλά και μεταδόσεων στο Euronews θεωρούμε ότι είναι από τα πιο έμπιστα μέσα για τους Ευρωπαίους και δίνουν πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ε, επίσης επισημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό και το δίκτυο ραδιοφώνου ε, με τρία νέα μέλη από την Εστονία, την Κύπρο και τη Σλοβακία το 2011. Έχουμε πλέον 22 επαγγελματικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και 8 πανεπιστημιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που, διαβιβάζουν, ε, που μεταδίδουν προγράμματα σε 21 γλώσσες και προσεγγίζουν πολλά εκατομμύρια πολίτες καθημερινά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να προωθούμε την πανευρωπαϊκή ε, συνιστόσα αυτού του ραδιοφωνικού συστήματος που είναι το πρώτο πανευρωπαϊκό σύστημα. Η Press Europe ε, είναι το πιο ε, πρόσφατο δίκτυο μαζικής ενημέρωσης. Προσφέρει ε, άρθρα, αναδημοσιεύσεις από διάφορες εφημερίδες, περιοδικά κλπ. Μεταφράζεται σε πολλές γλώσσες έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα φόρουμ. Έχει αυτό αυξήσει την ε, δημοφιλία του σε 500.000 ε, μοναδικές επισκέψεις ε, το 2011 και θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τις επισκέψεις το 2012. Επηρεάζει τον, τον διάλογο για τις δημόσιες πολιτικές, όπως για παράδειγμα τον διάλογο για την Συμφωνία Άκτα πολύ πρόσφατα. Χρειαζόμαστε επίσης και μια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Twitter, Facebook κλπ. Και, και άλλα έτσι ώστε και εκεί να συζητούνται τα ε, θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2011 ε, δημιουργήσαμε το δίκτυο ε, κοινωνικής ε, δικτύωσης της Κομισιόν. Εκεί συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι της τύπου της Κομισιόν από διάφορες γενικές διευθύνσεις, επιτρόπους και υπηρεσίες, έτσι ώστε να δίνεται μεγάλη δημοσιότητα σε διάφορα γεγονότα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, <clears throat> όπως η αιτήσια ομιλία του κ. Μπαρόσου. Ε, επίσης ε, θέλουμε να συμπεριλάβουμε ε, τη, την ε, κοινωνική δικτύωση στην υπηρεσιακή ομάδα τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα εφαρμόσουμε επίσης το πολιτικό πρόγραμμα του Κοινοβουλίου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε συνεργασία με τους δικούς σας εκπροσώπους τύπου στα κράτη-μέλη. Ε, έχουμε δεσμευθεί να συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητα ε, μέσα ε, και συνεργαζόμαστε με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας που έχει συγκεκριμένη έδρα για αυτό το θέμα. Ερχόμαστε σε Το κέντρο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει ε, η έδρα αυτή, το κέντρο αυτό έχει ξεκινήσει, ξεκίνησε τι δραστηριότητε του φέτο. Μία από τι δράσει που θα εφαρμόσει θα είναι ένα καλοκαιρινό σχολείο για δημοσιογράφου, επιχειρήσει ε, τύπου ε, και άλλου που καλύπτουν την ερευνητική δημοσιογραφία. Τώρα, το συμπέρασμά μου. θέλω να απευθύνω μια έκκληση σε εσά σε ό,τι αφορά τα αποθεματικά. Το αποθεματικό το οποίο τοποθετήσατε, στο οποίο τοποθετήσατε ένα τμήμα του προπολογισμού μας. Εμείς ακούσαμε τις συστάσεις σας και τις εφαρμόζουμε, τις υλοποιούμε και πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Αντίθετα με την αρχική μας θέση, κανονίσαμε να ξεκίνησει μία μελέτη βιωσιμότητας για το θέμα της ε, ε δράσης προετοιμασίας για την ερευνητική δημοσιογραφία σύμφωνα με τη δική σας τροπολογία του προπολογισμού 2012. Συνεπώ θα εφαρμοστεί και αυτή σα η επιθυμία. Περαιτέρω δε, βρήκαμε τρόπο να υλοποιήσουμε και το πιλωτικό πρόγραμμα ε, συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe, όχι αυτό το θέμα, το, το πρόγραμμα των υποδομών, είναι ε, ένα άλλο πρόγραμμα ε, που έχει στο κοπό να συνδέσει πολίτε μέσω των μέσων κοινωνική δικτύωση. Εσεί το, ζητήσατε, εσεί το ψηφίσατε και θα υλοποιηθεί από την Κομισιόν φέτο. Υπό το φω αυτών των ε, αυτών των δράσεων ζητώ από εσά να ε, ε, το, να απελευθερώσετε τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ που βρίσκονται στο απόθεμα που είχατε καθορίσει είναι πραγματικά ένα ποσό το οποίο το χρειαζόμαστε πολύ ε, και έχοντας ε, συζητήσει μαζί με πολλούς από εσά του τελευταίου μήνε, νομίζω μπορούμε να βρούμε μια συμφωνία που θα ικανοποιεί όλου. Ο τελικό στόχο τη Κομισιόν και του Κοινοβουλίου είναι ο ίδιο. Ε, η ε, Ευρώπη να κοινοποιεί και να δημοσιοποιεί τις πολιτικές της σε όλους τους πολίτες στην Ευρώπη έτσι ώστε να αυξηθεί η δημοκρατική συμμετοχή και να συνειδητοποιήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες τα δικαιώματά τους. Θα πρέπει η επικοινωνική πολιτική της Ευρώπης να ξεκινήσει σήμερα, όχι αύριο. Ε, ήδη έχουμε μπει, είμαστε σχεδόν στο Μάρτιο του 2012. Μόνο αν αρχίσουμε από τώρα θα μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για το ε, Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013 και το έτος των Ευρωπαϊκών Εκλογών 2014. Μην ξεχνάμε άλλωστε ε, ότι έχουμε το, τις δραστηριότητες για φέτος, να πέντε έτη ε, του Εράσμου, το Ευρωπαϊκό Έτος της Ενεργού Γύρανσης, ε, την ε, παρουσίαση της ε, νέας ε, κοινής αγροτικής πολιτικής κλπ, Όλα αυτά θα πρέπει να καλυφθούν με περιορισμένους πόρους που διαθέτουμε. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε να μας υποστηρίξετε. Δεδομένων των πόρων που διαθέτουμε και με τη δική σας συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Πόλγια. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα, κάτι που δεν περίμενα, ότι θέσατε ιδιαίτερη έμφαση στην διαθεσμική συνεργασία και πρέπει να σας πω ότι ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια δεν είχε πάει αυτό πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα που ένα μεγάλο μέρος των λόγων σας είχε θέσει ακριβώς στο επίκεντρό του την διαθεσμική συνεργασία. Δεν μπορούμε να προετοιμάσουμε μια προεκλογική εξατία αν δεν συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα. Θέλουν λοιπόν οι συνάδελφοι να έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν την εκλογή, τις εκλογές αυτές για τους πολίτες. Και η Κομισιόν η οποία εκλέγεται από εμά θα πρέπει να είναι και αυτή σε επίγνωση ότι υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Σας ευχαριστώ λοιπόν γιατί ήταν πολύ θετικό ότι αναφερθήκατε στο θέμα αυτό εκπεφρασμένα. Με την κυρία Ποδηματά και τον κύριο Καράς που είναι οι νέοι υπεύθυνοι αντιπρόεδροι πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια πραγματική πολιτική επικοινωνία και αυτό πρέπει να γίνει πραγματικότητα μέχρι το καλοκαίρι. Δεν πρέπει να περιμένει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από μόνο του παθητικά να γίνει κάτι. Πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο δράση και έχουμε ζητήσει από την κυρία Λαού η οποία είναι υπεύθυνη για τα θέματα επικοινωνίας να εφαρμόσει αυτό το σχέδιο επικοινωνίας. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά εν κενό αέρας. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση, δεν είμαστε αντίπαλοι, εργαζόμαστε για τον ίδιο στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση και για το μέλλον να έχει μια καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες, πάνω απ' όλα με τους νέους Ευρωπαίους πολίτες, να ξέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες γιατί θα πρέπει να δεσμευτούν και να αγωνιστούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαίρομαι λοιπόν και πάλι, όπως σας είπα, γιατί αναφερθήκατε για το κανάλι EPS και θέλω να σας υπενθυμίσω, πολλοί συνάδελφοι θυμούνται την ε, υπόθεση των ευρωπαϊκών χώρων, των αντιπροσωπιών της Κομισιόν και του Κοινοβουλίου να συνεργάζονται στις πρωτεύουσε δηλαδή των στις πρωτεύουσε των κρατών μελών και να έχουν και κοινέ δραστηριότητες, να υπάρξει μια κοινή οργάνωση ενεργειών. Πρέπει όμως να γίνει μια συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών και αυτό μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Και λέω και πάλι καλά τα λόγια, αλλά θα πρέπει να έχουμε και έργα. Και επίσης εντυπωσιάζομαι λιγάκι, διότι από τη δική μου την ε, πρακτική το Europe Direct δουλεύει πολύ καλά. Τουλάχιστον στη δική μου εκλογική περιφέρεια εργάζεται θαυμάσια. Μπορεί αλλού να μην εργάζεται να μην εργάζεται καλά. Αλλά το Europe Direct δεν είναι μονάχα φερέφωνο της ε, Κομισιόν. Είναι ο εκπρόσωπος όλων των θεσμικών οργάνων, οπότε περιλαμβάνει και το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Επομένως θα έχουν τη δυνατότητα οι βουλευτές να χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για να έχουν μεγαλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες τους. Επομένως νομίζω ότι όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμο να τα έχετε υπόψη σας. Είναι απαραίτητο να δώσουμε έμφαση στη διαθεσμική συνεργασία και το γεγονός ότι το αναφέρατε αυτό πολλές φορές στην παρέμβασή σας χαίρομαι γιατί θα ανατείλει μια νέα εποχή διαθεσμικής συνεργασίας. Η κυρία Καμεφέλντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Πάουγκερ για τις παρατηρήσεις του. Νομίζω ότι αυτά που ελέγχθηκαν για την διαθεσμική συνεργασία από την Προεδρό μας είναι πράγματα τα οποία τα υποστηρίζω απόλυτα. Όλοι περιμένουμε να ξεκινήσει μια νέα εποχή με εσάς επικεφαλής της επικοινωνίας. Ξέρουμε ότι στο παρελθόν ότι το Κοινοβούλιο πολλές φορές ενοχλήθηκε και εξοργίστηκε για την έλλειψη συνεργασίας. Ελπίζω λοιπόν θα μπορέσετε να επιλύσετε αυτά τα προβλήματα. Ένα παράδειγμα του πώς δεν θα πρέπει να συνεργαζόμαστε και ένα παράδειγμα του πώς θα μπορούσαμε να εργαζόμαστε καλύτερα είναι ακριβώς η διαθεσμική συνεργασία. Δεν είναι θέμα περιεχομένου, είναι ο, το θέμα που η Κομισιόν έχει ξεκινήσει διάφορες ενέργειες και τις έχει προωθήσει, μπορεί να έχουν σωστό περιεχόμενο, αλλά δεν έχει διαβουλευτεί καθόλου μαζί μας, δεν έχει ζητήσει τη γνώμη μας. Ελπίζω ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει στο μέλλον και νομίζω ότι τα λόγια σας δίνουν πράγματι ένα μήνυμα ότι η κατάσταση θα τροποποιηθεί. Θα ήθελα σχετικά να σας θέσω και ένα ερώτημα. Μιλήσατε για 4,5 εκατομμύρια στα μέσα για την επικοινωνία. Δεν έχω απέξω και ανακατοτά τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κεφάλι μου. Αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς θα σκεφτόσαστε να κατανείμετε αυτά τα 4,5 εκατομμύρια στις διάφορες ενέργειες και αυτό θα ήταν πολύ σημαντικό και για μας να το ξέρουμε πού θα θέσετε έμφαση, πού θα θέσετε το βάρος για τα κονδύλια αυτά. Κάτι άλλο το οποίο χαίρομαι είναι αυτά που είπατε και για τον ερευνητικό, την ερευνητική δημοσιογραφία. Είναι πάρα πολύ σημαντική η μορφή αυτή δημοσιογραφίας αλλά και εμείς είμαστε μεταξύ των θυμάτων μέσα σε εισαγωγικά αυτής της μορφής δημοσιογραφίας. Είναι σίγουρα ένας τρόπος να έρθουμε σε πιο να έρθει η Ευρώπη σε πιο στενή επαφή με το έργο του Κοινοβουλίου αλλά και της Κομισιόν και αυτό είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε στο προσκήνιο την Ευρώπη και το ίδιο ισχύει με τη συνεργασία αυτή που έχετε ξεκινήσει με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης. Αυτό σίγουρα ανταποκρίνεται στις αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι είναι ένα θετικό μήνυμα και μια θετική προσέγγιση και ελπίζω ότι θα μπορέσουν όλα αυτά να προχωρήσουν λίγο περισσότερο θα ήθελα όμως να μου απαντήσετε εφόσον μπορείτε για την κατανομή των ε, κονδυλίων γιατί τα κονδύλια αυτά δείχνουν ακριβώς και που στην πραγματικότητα θα τεθεί το μεγαλύτερο βάρος. Ευχαριστώ λέει και η Πρόεδρος. Κυρία Μακλάρκιν. Ευχαριστώ κύριε θα σας ευχαριστώ για την νέα ε, ε, θέση τι δύσκολο έργο που έχετε λάβει ιδίω με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη χώρα μου. Και ελπίζω να τα καταφέρετε να τους πείσετε για τα ωφέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή έχετε και αυτό το θέμα με το Ευρωπαϊκό Γραφείο το Επικοινωνίας, ε, το οποίο είναι 52 εκατομμύρια ευρώ των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην περιφέρειά μου, δεν γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τα ε, γεγονότα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει να φαίνεται ότι είναι ισορροπημένα τα πράγματα. Εμείς συνήθως ε, πιέζουμε μία ε, γραμμή και είναι πάντα προκατηλημένη. Θέλετε να δούμε και το ποιος είναι υπέλογο σε ποιον, αλλά πώς θα διασφαλίσουμε ότι είναι αμφίδρομη συζήτηση και δεν θα είναι μόνο μονόπλευρη. Επίσης ήθελα να ξέρω και να δω αν μπορείτε να μου το εξηγήσετε. Όταν λέτε ότι υποστηρίζετε δέκτια μέσων ενυπέρωσης και ότι έχετε ανεξάρτητους σταθμού, πώς είναι δυνατόν να είναι ανεξάρτητοι όταν τους χρηματοδοτείτε υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Γιατί αλλιώς δημιουργείται ερωτηματικός προς την ανεξαρτησία τους. Και ιδίως όταν έχουμε σεμινάρια για ε, δημοσιογράφους, ιδίως ε, ρεπόρτερ που κάνουν έρευνα, ε, τι ε, στοιχεία πρέπει να μας δώσουν στη συνέχεια. Εδώ τι γίνεται με την ελευθερία του λόγου. Θα πρέπει βέβαια να είναι οι πολίτε όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένοι, αλλά να προστατεύουμε και την ελεύθερη δημοσιογραφία και τα ελεύθερα μέσα ενημέρωση. Είναι διτός ο δρόμος και αφενός ε, υπάρχει το μήνυμά σας ε, και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθούν να τα προωθήσουν. Αλλά εγώ θα ήθελα όταν οι πολίτες είναι ενημερωμένοι και τους έχετε δώσει την έμπνευση ε, να μάθουν περισσότερα πράγματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρουν και από πού θα πρέπει να μπορούν να αποτανθούν. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αφού τους ζητάμε να είναι πιο έμεσα βλεγμένοι, θα πρέπει να μπορούν και κάπου να ζητήσουν πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ντόρις και εγώ από τη δική μου πλευρά θέλω να ευχαριστήσω τον Γκρέγορη Πόλγιο. Και εγώ όπως και οι άλλοι θέλω να τον ευχαριστήσω για την θέληση που έδειξε για συνεργασία, κάτι το οποίο το υπογράμμισε ιδιαίτερα και νομίζω ότι γνωρίζει ότι αυτό ήταν το κύριο σημείο των επικρίσεών μας και των αντιπαραθέσεων που είχαμε με την Κομισιόν στο παρελθόν. Θέλω επίσης να τονίσω ότι εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι σε σχέση με τη συνεργασία των δύο θεσμικών οργάνων θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη ισότητα και ισοτιμία των τριών κυρίων θεσμικών οργάνων και επομένως θα πρέπει να υπάρχει ισότιμη και ειλικρινής συνεργασία και από αυτά που είπε ο κύριος Πόλγκερ σήμερα νομίζω ότι το μήνυμα έχει φτάσει στον αποδέκτη του. Και θα ήθελα τώρα να αναφερθώ σε αυτά που είπε η κυρία Μακλάρκεν. Για μένα είναι πραγματικά πολύ διαφορετική η προπαγάνδα από την επικοινωνία. Όταν μιλάμε για επικοινωνιακή στρατηγική, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι αυτό δεν θα πρέπει να αφορά μονομερή προπαγάνδα ή να παρουσιάσει μόνο τις θετικές ή τις αρνητικές πλευρές μιας ενέργειας, αλλά πρόκειται για να δημιουργήσει ένα πολιτικό διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των πολιτών. Δεν ξέρω τι θα προκύψει καταρχήν από κάτι τέτοιο. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν τη σωστή πληροφόρηση και να ε, διαμορφώσουν τη δική τους άποψη. Αυτό είναι για μένα επικοινωνία χωρίς να υπάρχει κάποιο προσδιορισμένο αποτέλεσμα Γι' αυτό είναι ουσιαστικά μια προσφορά προς τους πολίτες για μια πολιτική αντιπαράθεση και συζήτηση. Οι πολίτες δεν θα είναι ικανοποιημένοι αν θεωρούν ότι απλώς εμείς τους πετάμε έτοιμο φαΐ, ότι είναι μια προπεγάνδα, κάτι το οποίο δεν είναι προς το δικό τους συμφέρον. Θα πρέπει να καταλαβαίνω ότι αυτό που γίνεται είναι μια διαδικασία που τους εμπλέκει. Μπορεί μερικές φορές αυτές οι απόψεις που διατυπώνει οι πολίτες να μην μας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η δημοκρατία. Αυτό πρέπει να σημαίνει ο διάλογος, να τους ζητούμε να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και να έχουμε και τη γνώμη τους για το μέλλον της Ευρώπης. Και ένα ακόμα τελευταίο σχόλιο θέλω να κάνω. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε μία συζήτηση για την ε, συμφωνία για τα δημοσιονομικά και μία ενδεχόμενη συνέλευση όπως παλιά με την ε, συνταγματική συνθήκη ώστε να έχει τη δυνατότητα το Κοινοβούλιο να κάνει ακουστή τη γνώμη του για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να ζητήσω και από την Κομισιόν ότι να γνωρίζει ότι αυτό σίγουρα θα είναι προς το κοινό συμφέρον μας, ιδίως εν ώψη των μελλοντικών ευρωεκλογών. Αν θέλουμε να παροτρύνουμε τους πολίτες να κατέβουν στις εκλογές, θα πρέπει να έχουμε κάτι να τους πούμε. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στην υπόλοιπη νομοθετική περίοδο το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνει σαφές προς τους πολίτες ότι έχει αρμοδιότητες και τους τις χρησιμοποιεί και μόνο έτσι θα πει στους πολίτες να έρθουν στις κάλπες. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι μονάχα απαραίτητο να λέμε για μεγάλες επιτυχίες, αλλά ένα παράδειγμα είναι το, η νομοθεσία του Six το εξαμερές αυτό νομοθέτημα, δεν θα υπήρχε χωρίς το Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε λοιπόν απλώ να πούμε ότι είμαστε οι μεγάλοι υπέρμαχοι τη δημοκρατία ή οι αγωνιστέ των πολιτών και μόνο, αλλά έχουμε σε ορισμένε συγκεκριμένε ενέργειε καταφέρει κάποια πράγματα. Πολλέ φορέ έρχονται ομάδε επισκεπτών στο Στρασβούργο και όταν του εξηγούμε τι έκανε το Κοινοβούλιο, τότε πραγματικά νιώθουν ότι κάτι έχουν καταλάβει, ότι κάτι αρχίζουν να κατανοούν από το πώ δουλεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περάσει κάποιες απόψεις και έχει επικρατήσει του Συμβουλίου, η Κομισιόν πάντα πρέπει να λέει ότι εμείς κάνουμε μεν τις προτάσεις, αλλά η νομοθετική διαδικασία περνά από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και είναι τα δύο σχέδια της νομοθετικής εξουσίας που θα πρέπει να πάρουν την τελική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν η Κομισιόν και το ε, Κοινοβούλιο να συνεργαστούμε και η κυρία Επίτροπος να καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνη της η οποία εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει και το Κοινοβούλιο να είναι παρό. Κύριε Βεζιά. Oui, merci Madame la Présidente, merci euh, Monsieur, Monsieur le Directeur. Euh, je vais aller dans le même Θα μιλήσω ε, με παρόμοιο τρόπο με τους προηγούμενους συναδέλφους. Ε, βέβαια έχω την εντύπωση ότι ε, ότι ότι δεν γίνεται κάποιος διάλογος για την ε, πολιτική επικοινωνία στην επικοινωνική πολιτική της Κομισιόν, ότι αποφασίζεται εκ των άνω και επιβάλλεται προς τα κάτω. Ε, δεν καταλαβαίνω πώς λαμβάνονται υπόψη οι πολίτες και δεν καταλαβαίνω και πολύ καλά την πολιτική για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν πάρα πολλέ σελίδε για τα ευρωπαϊκά θέματα εκεί, αλλά δεν είναι σελίδε διαλόγου, είναι σελίδε μόνο ενημερωτικέ. Τα δίκτυα, ε, η κοινωνική, δικτύωση ε, δεν γίνεται για αυτό το λόγο, για να ενημερώνονται οι αναγνώστες. Η ενημέρωση δεν βοηθάει σε τίποτα. Χρειάζεται διάλογο. Λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Να σας δώσω ένα Παράδειγμα, ψηφίσαμε σήμερα το πρωί για την Ευρώπη των πολιτών. Είναι ένα προσφυλές μου θέμα. Ε, εγώ ζήτησα μάλιστα να αλλάξουμε και το όνομα. Αλλά εντάξει, δεν συμφωνήσα μαζί μου ΑΛΦΗ, αλλά εν πάση περιπτώσει ε, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που τα άλλα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θέλουν να ακούσουν αυτό που λέει το Κοινοβούλιο. Γιατί ο καθένα έχει μπλοκαριστεί στην δική του, ε, στο δικό τρόπο να βλέπει τα πράγματα. Δεν επικοινωνούμε με τον πολίτη. Και δεδομένου ότι ε, το 2014 έχουμε ε, και εκλογές, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πιο σοβαρό λόγο, πιο δυνατό λόγο για το πώς θέλουμε να είναι το έτος του Ευρωπαϊκού Πολίτη. Ε, σήμερα το πρωί αυξήσαμε τον προπολογισμό στα 5 εκατομμύρια. Εδώ και πολύ καιρό ε, λέτε ότι χρειάζονται, ότι δεν χρειάζεται να αυξήσουμε τι ε, πιστώσει, γιατί υπάρχουν ε, πιστώσει από αλλού, δεν ξέρω από πού είναι αυτέ τι πιστώσει. έχω ρωτήσει, ε, δεν μου έχει λεχθεί, δεν μου έχει δοθεί απάντηση, θα ήθελα να ακούσω. Ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα, έτσι. δεν περιμένω μια απάντηση σήμερα, αλλά είναι ένα παράδειγμα για να σας δείξω ότι δεν δουλεύουμε σωστά. Και υπάρχουν και άλλα τέτοια παραδείγματα. Μετά, για το θέμα του αποθεματικού, για το, στο οποίο αναφερθήκατε. Και εκεί χαρακτηριστικά ε, ε βρισκόμαστε στο ίδιο σχήματο. σχήματο. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε αυτά τα ποσά σε αποθεματικό όχι για να τα χρησιμοποιήσει η Κομισιόν για να φτιάξει τη δική της εικόνα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο project πίσω από αυτά που είναι η Πανευρωπαϊκή Τηλεόραση η απάντηση της Κομισιόν, αν κατάλαβα καλά, ε, ήταν να θέσει το περιθώριο αυτό το project ε, και να χρησιμοποιήσει τα ίδια ποσά ε, με βάση τη, δική, τη δική της επικοινωνιακή πολιτική. Εγώ έτσι δεν θα απελευθερώνω το αποθεματικό. Όχι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και η Πρόεδρος. Να προσθέσω κάτι ακόμα κι εγώ. Αυτό που μου άρεσε ακριβώς ήταν το θέμα της Press Europe που ανέφερε ο Σπόλγερ. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το διεθνή τύπο, αλλά είναι πολύ χρήσιμο οι Ευρωπαίοι πολίτες κάθε εθνικότητος να δουν ότι αυτά τα στοιχεία του τύπου μπορούν να μεταφράζονται τουλάχιστον σε 10 γλώσσες να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν αυτά τα οποία τυπώνονται σε εφημερίδες για τα θέματα που τους απασχολούν στη χώρα τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση των χωρών της Ευρώπης και θέλω να σας συγχαρώ για το γεγονός ότι υποστηρίζετε το Press Europe και είναι μια πολύ καλή ιδέα. Κάτι ακόμα όμως, ένα ερώτημα. Είπατε ότι θα εκπνεύσει το πρόγραμμα Europe Direct και αναρωτιέστε αν θα πρέπει να κάνετε μια προσπάθεια να να σκεφτείτε για την ανανέωσή του και να κάνετε τον αντίστοιχο διαγωνισμό. Εμείς το έχουμε επενέσει αυτό το πρόγραμμα, σας λέω τουλάχιστον στη δική μου χώρα θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ σημαντικό για μας λοιπόν να συνεχίσει το Europe Direct ως πρόγραμμα. Ένα παράδειγμα μας αναφέρθηκε η κυρία Βερζιά στο έτος των πολιτών. Είναι ένα χρόνο το 2013 πριν από τις ευρωεκλογέ. Θα πρέπει να έχουμε προγράμματα φάρους τα οποία θα μπορέσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών. Ή το βραβείο Λουξ, παραδείγματος χάρη, για τον κινηματογράφο. Πριν από την απονομή του βραβείου εδώ, τον Νοέμβριο πέρσι, είχαμε πει να κάνουμε μια εβδομάδα κινηματογράφου. Με τις ε, επιλεγμένες ταινίε και κάποιες ακόμα. Σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης και σε άλλες ε, ε, περιπτώσεις, σε πόλεις όπου έχουμε γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να κάνουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και θα δειχνόντουσαν λοιπόν τα ταινία αυτά σε ειδικέ αίθουσε οι οποίες θα τα προβάλλανε δωρεάν. Αυτό ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Χρειαζόμασταν μια υποστήριξη από εσά. Όχι να μα πάρει το ραδιολούξ, το οποίο είναι δική μα ιδέα, αλλά να συνεργαστεί μαζί μα η Κομισιόν για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η δυνατότητα μετά από την προβολή των ταινιών αυτών να γίνουν συζητήσει. Κάτι που θα πολλαπλασίασε και το αποτέλεσμά του. Είχαμε τη δυνατότητα έτσι να συζητήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι ποτέ δεν θα πήγαιναν σε μια εκδήλωση για την Ευρώπη να συζητήσουν για αυτά τα θέματα. Όχι ανθρώπου που του ενδιαφέρει η επικαιρότητα, ανθρώπου που είναι κινηματογραφόφιλοι. Να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τα άτομα αυτά για την Ευρώπη. Είναι ένα νέο σύγχρονο μέσο με το οποίο μπορούμε να πλησιάσουμε τους πολίτες. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε τη βοήθεια της Κομισιόν αν πάρετε τις απαραίτητες αποφάσεις θα μπορούσε να γίνει αυτό το 2012 ήδη. Θέλουμε λοιπόν τη βοήθειά σας για τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα και αυτό είναι παράδειγμα ιδεών που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν το έτος 2013. Από κοινού θα πρέπει στην επόμενη συνάντηση που γίνεται μέσα στα πλαίσια της ομάδας επικοινωνίας να συζητήσουμε ακριβώς ποιες είναι οι συγκεκριμένες και μεμονωμένες ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε τον επόμενο χρόνο και να δούμε πώς θα κατανοούμε τους πόρους στον προϋπολογισμό που έχουμε για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να σας δώσω το λόγο λοιπόν κύριε Πόλγκερ για να απαντήσετε τώρα. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη για τις ερωτήσεις τους και τις παρατηρήσεις τους. Καταρχάς, για το αποθεματικό. Πρόκειται για ένα αποθεματικό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ σε μία γραμμή προϋπολογισμού, τη γραμμή για τα ε, μέσα δικτύωσης που περιλαμβάνει το Euronews, το Euronet και το Press Europe. Πρόκειται για προγράμματα τα οποία η Επιτροπή σας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη υποστηρίζει. Για να μπορέσουμε να πληρώσουμε πλήρως αυτό που χρωστάμε σε αυτά τα δίκτυα φέτος, χρειαζόμαστε αυτά τα κονδύλια. Είναι συμβατική υποχρέωση. Ως διαχειριστή, βεβαίω εγώ ενδιαφέρομαι ε, για το σεβασμό των συμβατικών υποχρεώσεων και μάλιστα εγκαίρω. διότι αν δεν χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια φέτος θα χαθούν. Όλα αυτά τα κονδύλια θα μας επιτρέψουν επίση να ενισχύσουμε και την γλωσσική κάλυψη του Euronews. Για παράδειγμα, στις χώρες προγράμματος, ε, διότι βιώνουμε και χαλεπούς οικονομικούς καιρούς, στις χώρες λοιπόν προγράμματος, όπου μεταδίδεται το Euronews ε, μέσω ε, των δημοσίων δικτύων στην εθνική γλώσσα, αυτές οι μεταδόσεις αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές πιέσεις. Η συγκεκριμένη λοιπόν γλωσσική εκδοχή του Euronews μπορεί να μην χρηματοδοτείται πλέον από τη δημόσια τηλεόραση. Αυτό ισχύει για παράδειγμα για την Πορτογαλία, όπου το Πορτογαλικό Κοινοβούλιο ανησυχεί ιδιαίτερα και φοβάται ότι θα σταματήσει η μετάδοση στην πορτογαλική γλώσσα, διότι πλέον δεν δίνονται τα απαραίτητα κονδύλια για να χρηματοδοτηθεί η γλωσσική εκδοχή στα πορτογαλικά. Εάν έχουμε τα κονδύλια αυτά τα οποία είναι διαθέσιμα στο αποθεματικό αυτό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ευρώ θα μπορούμε ε, επιμονή μου βάσεως πλέον για την προγραμματική περίοδο που διανύουμε τώρα, έχουμε φτάσει βέβαια στο τέλος της διαδρομής, αλλά ε, θα ξανάρθουμε στην αρχή ε, και στην κορυφή και οι χώρες αυτές δεν θα είναι πλέον χώρες προγράμματος εάν φτάσουμε εκεί. Βρισκόμαστε λοιπόν στον πάτο και επειδή ακριβώ βιώνουμε χαλεπού καιρού, θέλουμε να βοηθήσουμε τι χώρε αυτέ με διάφορου τρόπου. Και ένα από του τρόπου με του οποίου μπορούμε να τι βοηθήσουμε είναι να διατηρήσουμε τη δική του γλωσσική εκδοχή ε, στη μετάδοση του Euronews. Ε, πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Και δεν θα μπορέσει να γίνει αυτό χωρί αυτό το αποθεματικό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα λοιπόν του πώ θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Απαντώ και πάλι στην κυρία Κάμεβελτ. Ναι. Η δημοσιογραφία και μάλιστα το έργο των ρεπόρτερ είναι ένα τομέα ο οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό από πολλά μέλη τη συγκεκριμένη επιτροπή. Και γι' αυτό ακριβώ ε, αναλάβαμε και τι δύο συγκεκριμένε δραστηριότητε. Αυτή η οποία σα ανέφερα του Πανεπιστημίου τη Φλωρεντία, όπου υπάρχει συνεργασία για την ακαδημαϊκή πτυχή της δημοσιογραφίας ε, και η άλλη πτυχή είναι ε, τα σεμινάρια αυτά τα οποία σας ανέφερα και θα εφαρμόσουμε, αντίθετα με τα όσα πιστεύουμε, την προπαρασκευαστική δράση που ψήφισε η Επιτροπή σας για το 2012. Θα εφαρμοστεί λοιπόν αυτόν. Είναι μια συγκεκριμένη δράση για την ε, ερευνητική δημοσιογραφία και θα δούμε πώς ε, μπορούν να υποστηριχθούν συγκεκριμένα προγράμματα για την διερευνητική αυτή δημοσιογραφία μέσω μιας μελέτης σκοπιμότητας. Συμφωνώ και με την κυρία Μακλάρκεν και με την κυρία Τρίπελ ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναζητούν οι πολίτες και μάλιστα εύκολη πρόσβαση, ε, αμερόληπτη οι πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζονται ουδέτερες ε, ως γεγονότα. Εμείς ε, στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας δεν θεωρούμε ότι είμαστε Υπουργείο Επικοινωνίας ε, παλιού τύπου. Είμαστε εκεί για να σας αναφέρουμε πως έχουν τα γεγονότα και μάλιστα να τα αναφέρουμε με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό και προσιτό τρόπο και μάλιστα μερόληπτα. Υπάρχουν αρκετά εργαλεία στη διάθεσή μας για να γίνεται αυτό. Υπάρχουν χιλιάδες πολίτες κάθε χρόνο οι οποίοι χρησιμοποιούν την υπηρεσία Europe Direct. Εγώ επισκέφθηκα την υπηρεσία την περασμένη εβδομάδα και είναι εκπληκτικό αυτό που κάνουν. Είναι εδώ στις Βρυξέλλες, στο κέντρο, είναι πολύ πιο ανθρώπινα τα πράγματα από αυτά που έχουμε στο νου μας. Δεν είναι ένα κέντρο ε, τηλεφωνικό, είναι ένα ε, υψηλής τεχνολογίας κέντρο. Ε, έχουμε νέους ανθρώπους, όταν ε, λέω νέους εννοώ στα 20 τους, πολύ καλά καταρτισμένους για την Ευρώπη, όλοι έχουν μάστερ σε ευρωπαϊκές σπουδές, οι οποίοι μιλούν και τις 23 γλώσσες, συνάντησα έναν ε, νεαρό ο οποίος είναι ειδικό ε, στις πληροφορίες για τα ερευνητικά προγράμματα, ο οποίος απαντά ερωτήσεις στα Ιρλανδικά. Όλοι μιλούν τουλάχιστον τρεις γλώσσες και αυτοί οι άνθρωποι ε, υπάρχει ένας δωρεάν τηλεφωνικός αριθμός, οι πολίτες μπορούν να τηλεφωνήσουν σε αυτόν τον αριθμό και τηλεφωνούν και μπορούν να ζητήσουν απευθείας πληροφορίες και να τους απαντηθούν αμέσως ή αν είναι πιο περίπλοκο το ερώτημα, τους ε, παραπέμπουν στην κατάλληλη πηγή. Πέρσι είχαμε 70 με 80 χιλιάδες τηλεφωνικές κλήσεις από πολίτες ε, από όλη την Ευρώπη σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Διατίθενται όλε οι γλώσσε Ευρωπαϊκή Ένωση και όπως σας είπα, λαμβάνουν απάντηση απευθείας ε, από τον άνθρωπο με τον οποίο συνομιλούν στο τηλέφωνο. Ή υπάρχει και μια ε, υπηρεσία διαδικτύου, υπάρχουν αρκετέ ερωτήσει που φτάνουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι πολίτε που θέτουν ερωτήσει λαμβάνουν απάντηση εντό τριών ημερών στη γλώσσα του μέσω του κέντρου Europe Direct. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο. Και επειδή η κυρία Βερζιά αναφέρθηκε στην ε, ε, επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω, μία από τις υπηρεσίες που αναπτύσσει το Europe Direct είναι ένα τμήμα ε, chat, συνομιλία στο διαδίκτυο, όπου κάποιος ε, μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία μέσω διαλόγου στο διαδίκτυο. Και αυτό φυσικά είναι από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Μπαίνω, κάθομαι σε ένα τραπέζι και λαμβάνω απάντηση από το Europe Direct. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα παραδείγματα που καταδεικνύει πώς οι πληροφορίες είναι στη διάθεση του πολίτη. Όσον αφορά τώρα την ισορροπημένη συζήτηση και την ανάγκη ανεξαρτησίας, ναι βεβαίως το υποστηρίζουμε αυτό. Δεν υποστηρίζουμε το Euronews. Το Euronet, το Press Europe, με όλους αυτούς έχουμε συμβάσεις. Και όλες οι συμβάσεις περιλαμβάνουν μία ρήτρα που λέει ότι ε, είναι υπεύθυνη για τα όσα γράφονται. Υπάρχει ελευθερία ε, ως προς το τι γράφεται. Από εκεί και πέρα τα θέματα και τα προγράμματα είναι ευρωπαϊκά ε, ή έχουν σχέση με την Ευρώπη. Αλλά Οι τηλεοπτικοί σταθμοί είναι αυτοί που επιλέγουν ε, τι ακριβώς θα προβάλλουν. Υπάρχει απόλυτη ελευθερία από αυτού και νομίζω ότι ένα από τα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε για κάποια από τα μέλη του Euronet είναι το European Press Review. Ε, αυτό είναι εξορισμού ανεξάρτητο μέσο διότι γίνεται μια προφορική σύνοψη σε ραδιοφωνικά προγράμματα του τι περιλαμβάνεται στον ευρωπαϊκό τύπο καθημερινός. Ε, αυτό είναι ουσιαστικά αντικειμενική δημοσιογραφία. και είναι ένας καλός τρόπος να ενημερώνουμε τους καθημερινούς πολίτες για το τι συμβαίνει στις χώρες ε, στην Ευρώπη. Τώρα να δω τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν κατέχει κανείς ακόμα και μάλλον δεν θα πρέπει κανείς να το κατέχει, διότι εξορισμού είναι μια έκφραση ελευθερίας και κάποιες από τις μεγάλες επιχειρήσεις που προσπάθησαν ε, να τελειοποιήσουν τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ε, με μονόπλευρο τρόπο απέτυχαν παταγωδός και γύρισε και τους χτύπησε μπούμεραγκ. Θα πρέπει κάποιο να είναι πλήρω μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να συνδιαλέγεται με τους πολίτες στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Αυτή είναι μια τεχνική την οποία θα πρέπει να αναπτύξουμε. απαιτεί κάποιο βαθμό επαγγελματισμού. Όλοι μαθαίνουν βαθμιδών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά νομίζω ότι αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε και είναι πολύ θετικό χάρη σε εσά φέτο, είναι να εφαρμόσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο προώθησε η Επιτροπή σα για την, ε, ε, ε, το, την Ευρώπη στο διαδίκτυο. Αυτό θα γίνει με αποκεντρωμένο τρόπο μέσω των μονίμων αντιπροσωπιών και των γραφείων ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα μα δώσει πολύτιμη ε, εμπειρογνωμοσύνη επί του θέματος. Τώρα, όσον αφορά το ευρωπαϊκό έτος, ε, κυρία Βερζιά, Βεβαίω και ακούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο συνομοθέτη. Εμεί προτείνουμε, εσεί αποφασίζετε. Δεν είναι θέμα μόνο του κατά πόσον τίνουμε δίκονου. Εσεί είστε ο, ο, ο νομοθέτης, εσείς έχετε αυτό το ρόλο και εμεί κάνουμε προτάσει για να τι επεξεργαστείτε και να τι βελτιώσετε. Έτσι λειτουργεί το θεσμικό σύστημα. Νομίζω ότι με αυτά κάλυψα τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις, κυρία Πρόεδρε. Αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένο, κυρία Περαμπαραδού, σας ευχαριστώ. Μίλησατε για τη σημασία των ε, τηλεοπτικών ε, μέσων. Είναι ε, μέσα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν πάρα πολλούς πολίτες, αλλά η σωστή στρατηγική είναι να έχετε μια τηλεόραση δικιά μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι το Euronews ή είναι καλύτερο να δίνουμε προϊόντα, επικοινωνιακά προϊόντα, φιλμάκια, υλικό στα, το, στα γενικά μέσα ενημέρωσης τα οποία έχουν πρόσβαση στους πολίτες. Πόσοι κοιτάζουν τα Euronews, μόνο αυτοί που είναι οι δήμονες και ενδιαφέρονται για την Ευρώπη. Μα ο στόχος σας θα πρέπει να είναι να Παρακινήστε το ενδιαφέρον άλλων πολιτών που δεν ξέρουν τίποτα για την Ευρώπη. Ίσως μια άλλη στρατηγική θα ήταν να έχετε συμβάσεις με, μεγάλες, με μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια ευρεία διάδοσης και τα οποία μπορούν να συνεργάζονται μαζί σας με τα στοιχεία που, σας, που δίνετε για να μπορέσουν να ε, προσελκύσουν το ενδιαφέρον των πολιτών πέραν από αυτών οι οποίοι είναι ήδη μοιημένοι. Κύριε Μπεναραμπατού, Μπεναρά προτού απαντήσετε, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πει στα κανάλια τι θα δείξουν και τι δεν θα δείξουν. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε μια έκκληση στα κανάλια να δείχνουν περισσότερο το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ήδη στα μεγάλα, στα μεγάλα γερμανικά κανάλια υπάρχουν προγράμματα για την Ευρώπη, αλλά δεν είναι επαρκή. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να τους επιβάλλουμε κάτι τέτοιο, εκτός αν ο κ. Πόλγκερ έχει να μας προτείνει κάτι σχετικά. Βεβαίω λέει ο κ. Πόλγκερ. Τα μεγάλα εθνικά τηλεοπτικά κανάλια ασφαλώς έχουν κάποιο ρόλο να παίξουν είτε πρόκειται για κρατική τηλεόραση που έχει συγκεκριμένους ε, κανόνες ε, που μεταξύ αυτών μπορεί να είναι πολλές φορές και η κάλυψη των ευρωπαϊκών θεμάτων δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε ε, είτε είναι ιδιωτικά κανάλια το πλειονέκτημα τέτοιων συμφωνιών με τέτοιου είδους κανάλια είναι ότι μας δίνουν πρόσβαση σε ένα κοινό το οποίο ήδη υπάρχει. Η France 2 ας πούμε έχει 5 με 10 εκατομμύρια τηλεθεατές ημερησίως ε, στις ώρες αιχμής. Δεν είναι εύκολο κανείς να το φτιάξει αυτό από το μηδέν, ακόμα και αν το επιθυμεί. Αυτό που μπορούμε όμως να κάνουμε το Euronews είναι το εξής ο περιορισμός του Euronews μέχρι τώρα ήταν ότι το Euronews ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω δορυφόρου. Προφανώς αυτό ε, είναι αρκετά περιοριστικό διότι η δορυφορική τηλεόραση είναι ένας μόνο τρόπος να φτάσει, να φτάσει ε, το πρόγραμμα στα σπίτια των ε, πολιτών. Όμως τώρα το Euronews έχει περάσει στην καλωδιακή τηλεόραση. Σύντομα φτάνει η επίγεια ψηφιακή τηλεόραση όπου δεν έχει φτάσει ακόμα, μέσω της οποίας πολλοί ε, τηλεθετές θα έχουν πρόσβαση στο Euronews. Και στα κράτη-μέλη πολύ συχνά βλέπουμε, μάλλον όλο και πιο συχνά βλέπουμε, ε, ε η, ε, τα διάφορα κανάλια να αναμεταδίδουν για δύο ώρες για παράδειγμα ε, την εκπομπή του Euronews μέσα στο δικό της πρόγραμμα. Αυτό ασφαλώς είναι πολύ καλό και σίγουρα η κατάσταση βελτιώνεται. Η κυρία Κάμεβερτ. Θα ήθελα να πω και κάτι για αυτό το ερώτημα. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό και η Κομισιόν να δώσει έμφαση στο να γίνονται σεμινάρια και για τους δημοσιογράφους. Γιατί έχουμε ένα προϋπολογισμό για τα ευρωπαϊκά θέματα, γιατί θα πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες παραγωγικά σε τοπικούς δημοσιογράφους να ξέρουν κάτι περισσότερο για τα ευρωπαϊκά θέματα, να τους δώσουμε και κίνητρα να απασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα. Γιατί βλέπουμε παραγωγικά στα blog που λένε πράγματα που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα στην Ευρώπη. Είναι απαραίτητο λοιπόν όταν δουλεύουμε παραγωγικά με τα δημόσια ε, ραδιόφωνα να τους ε, παρακινήσουμε όχι να τα βάζουν όλα αυτά μονάχα σε μία εκπομπή αλλά να είναι κάτι το οποίο συζητάτε σε όλα τα επίπεδα γιατί στη Γερμανία όταν κάνουν μια συζήτηση για την Ευρώπη κλείνουν όλοι πανικόβλητοι τα ραδιόφωνά τους λοιπόν πρέπει στα κανονικά νέα και τις ενημερώσεις η Ευρώπη να περιλαμβάνεται και να υπάρχει λοιπόν μια πληροφόρηση για το τι γίνεται στην Ευρώπη και όχι να υπάρχει σε ένα γκέτο η Ευρώπη ή να υπάρχουν πολιτικά μαγαζίνα τα οποία έχουν μια κριτική αντιπαράθεση για την Ευρώπη. Να φτιάξουμε λοιπόν χώρους οι οποίοι να περιλαμβάνουν τα ευρωπαϊκά θέματα σε ένα προς ένα ευρύ κοινό, αλλά καταρχήν θα πρέπει να πείσουμε τους δημοσιογράφους πρώτον ότι κάνουμε χρήσιμη και σημαντική εργασία και μετά να την προβάλλουμε και αυτό είναι σημαντικό να προωθήσουμε τα σεμινάρια για τους τοπικούς αρχισυντάκτες και συντάκτες για να έχουν την απαραίτητη κατάρτιση για τα ευρωπαϊκά. Κάτι ακόμα θέλω να προσθέσω, λέει η Doris Πακ. Εδώ ε, το πρόβλημα είναι ότι συζητάμε κάτι, ψηφίζουμε σε πρώτη ανάγνωση, μετά πηγαίνει στο Συμβούλιο. Το Συμβούλιο χρονοτριβεί για να καταλήξει σε μία συμφωνία και σε τελική ανάλυση το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο αποφασίζει. Επομένως, το Κοινοβούλιο δεν έχει πολλές φορές τον τελικό λόγο και οι δημοσιογράφοι δεν καταλαβαίνουν πώς γίνεται αυτή η διαδικασία και επομένως δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία και να την παρουσιάσουν στους ακροατές τους. Αν δεν θέλει κανείς ένα ερώτημα να θέσει, θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον κύριο Πόλγκερ. Χαιρόμαστε για την παρουσία σας και πιστεύω ότι το γνωρίζουμε φυσικά και από τις δραστηριότητε του στο παρελθόν. Χαιρόμαστε που έχει αναλάβει αυτή την αρμοδιότητα. Ελπίζουμε ότι έχουμε μαζί σας ένα σημαντικό συνομιλητή και αυτά τα οποία αναφέρατε εδώ ε, μεγαλοφόνος η διαθεσμική συνεργασία είναι σημαντικά, χαιρόμαστε που τα αναφέρατε και θα εξετάσουμε πράγματι το θέμα της απελευθέρωσης του αποθεματικού όπως ζητήσατε γιατί εάν είναι σαφές ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τις κατάλληλες ενέργειες. Και πάλι σας ευχαριστώ και γεια σας. Μέχρι την επόμενη φορά. Okay. Jetzt kommen wir zum Punkt 12. Σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης προστασία των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο. Έκθεση πρωτοβουλία της κυρίας Σίλβια Κώστα. Σα δίνω αμέσω το λόγο Σίλβια. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα θέμα και καινοτόμο, διότι έχει λάβει μορφές ε, η ψηφιακή επικοινωνία και η χρήση των ψηφιακών μέσων από πλευρά ανελίκων, αλλά φυσικά έχουμε και νέα νομοθετικά μέσα και νέε προσεγγίσει, οι οποίε κατά την άποψή μου θα πρέπει να προαχθούν. Η συγκεκριμένη έκθεση ιδέα πρωτοβουλία απαντά στην έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, του 2011 για την εφαρμογή σύστασης ε, του Συμβουλίου του 1998 για τη μέθοδο ανταγωνιστικότητας του κλάδου και των ε, ο, οπτικοακουστικών υπηρεσιών, αλλά ήθελε και να είναι πιο ανταγωνιστικό ο τομέα ε, των οπτικοακουστικών μέσων, αλλά ταυτόχρονα να προστατεύονται και καταλήλω ε, οι ανήλικοι. Ε, από αυτό είχαμε μία σύστοση ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών του Δεκεμβρίου του 2006 ε, ως απάντηση για τα όσα συμβαίνουν στα οπτικοακουστικά μέσα και της διαδικτυακής ενημέρωσης. Αυτή είναι η πρώτη αναφορά που έχουμε στο θέμα αυτό. Στη σύσταση προβλεπόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τακτικά εκθέσεις για να δει κατά πόσον εφαρμόζεται αποτελεσματικά από πλευράς κρατών μελών αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής η νομοθεσία με στόχο ίσως και μια σχετική αναθεώρηση. Το πρώτο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω στην εκθεσή μου λοιπόν είναι να επαληθεύσουμε πώς άλλαξαν οι συνθήκες ε, χρήσης από πλευράς ανηλίκων των ψηφιακών δυνατοτήτων που τους προσφέρονται, που τους προσφέρουν φυσικά πολλές δυνατότητες αλλά φυσικά και νέους κινδύνους και ε, αυτό προκύπτει και από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από διαβούλευση με τα κράτη-μέλη. Σίγουρα δεν επαρκεί να υπάρχει μόνο νομικής φύσεως προσέγγισης παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές όπου δεν εγγυόμαστε την προστασία ή είναι λυπής η προστασία. Θέλουμε να έχουμε όμως μια πιο ολιστική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη και ε, τον ψηφιακό κόσμο ε, και ως μια μεγάλη ευκαιρία ε, για παιδεία, για αλληλεπίδραση, ε, ανάπτυξη δεξιοτήτων, αλλά φυσικά και ίσως μια ευκαιρία μεγαλύτερης έκφρασης μιας ψηφιακής υπηκότητας ε, να υπάρχει ενεργό συμμετοχή και δυνατότητα των ανηλίκων να αναπτυχθούν μέσω αυτής της διαδικασίας. Αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο έχει αλλάξει αρκετά στο τελευταίο διάστημα. Θα ήθελα απλώς να σας αναφέρω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ότι υπάρχει νομική βάση που επιτρέπει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η διάθεση να προχωρήσουμε λίγο περαιτέρω και να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη δράση. Ίσως, και αυτό επιτρέψτε μου να σας το προτείνω, να έχουμε και μια οδηγία που θα είναι ένα ενιαίο κείμενο και θα συλλέξει όλες τις διάφορες μορφές προστασίας, προώθησης, ε, και προστασία των δικαιωμάτων και έκφραση των δικαιωμάτων των ανηλίκων στο ψηφιακό κόσμο που αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτα σε διάφορε οδηγίε. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην οδηγία για τα οπτικοακουστικά μέσα που δεν αναφέρεται καθόλου στα ψηφιακά θέματα, στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στην διαδικτυακή τηλεόραση ε, ή την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο που αναφέρει μεν κάποια στοιχεία για την προστασία των ανηλίκων σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου ε, ή υπάρχει οδηγία που προβλέπει και διευρύνει θέματα προστασίας ανηλίκων και προβλέπει και κάποιες συγκεκριμένες ε, περαιτέρω συστάσεις ώστε να προστατεύουμε ε, και διαδικτυακά τους ανηλίκους και υπάρχει και οδηγία για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια του 2008 που είχε την δυνατότητα σταδιακής πρόσβασης βάσει ηλικίας και άλλων κριτηρίων που στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε ένα πολύ σημαντικό σύστημα αυτορύθμισης, το PEGI, ε, το οποίο είναι μία από τις πολύ καλές εφαρμογές, ένας κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος αναπτύχθηκε αυτόνομα από τον ακουστικό τομέα για να προστατεύουν, αλλά ταυτόχρονα να δίνουν και κάποιες υποδείξεις για την κατάλληλη ηλικία ε, και το ε, κατά πόσον είναι κατάλληλα κάποια ηλεκτρονικά παιχνίδια για ανηλίκους. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ε, ως πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη έκθεση ένα ε, πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το Safer Internet Programs ε, του 1999, το οποίο ανανεώθηκε και διαφοροποιήθηκε μέχρι και το 2013 και ελπίζω και θα το ζητήσω αυτό να χρηματοδοτηθεί εκ νέου μέσω του προγράμματος Connecting Europe στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Πάολγκερ προηγουμένως αλλά να υπάρχει και ιδιαίτερη προσοχή εντός αυτού του τόσου μεγάλου προγράμματος που θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τα θέματα του διαδικτύου διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις ιδιαιτερότητες του Safer Internet διότι το ασφαλέστερο διαδίκτυο κατ' εμέ είναι τα τρία στοιχεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να φροντίσουμε να τα προωθήσουμε περαιτέρω. Δηλαδή, αφενός, μια πρώτη γραμμή είναι να υπάρχει συντονισμός ε, όλων των γραμμών βοήθειας ε, σε όλη την Ευρώπη ε, που παρουσιάζονται από συγκεκριμένους οργανισμούς. Αυτό είναι πολύ μεγάλη κληρονομιά κάθε χώρας και να κυριαρχούν ε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεύτερον, όλοι οι ανήλικοι να έχουν ε, ε, ποιοτικέ διαδικτυακές υπηρεσίες και τρίτον, στο Safer Internet υπάρχει μεγαλύτερη μάχη κατά του παράνομου περιεχομένου ε, ή κατά, καταλα, κατάλληλου περιεχομένου για τους ανηλίκους και να προάγουμε τη συνεργασία μεταξύ του κλάδου, των μη κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και των δυνάμεων της τάξης. Ε, όλα αυτά φυσικά περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Ε, η, θα ήθελα να προτείνω τα εξής. Καταρχάς θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση και προσπάθησα ακριβώς αυτό να κάνω ε, και να ε, χωρίσω την έκθεσή μου σε τέσσερις άξονες. Καταρχάς να σκεφτούμε το όλο θέμα της διακυβέρνησης του θέματος αυτού και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ε, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα και τα κράτη-μέλη να βρουν εθνικά σημεία αναφοράς συντονισμού τα οποία ε, θα περιλαμβάνουν όλους τους ενδιαφερομένους ε, σε θέματα προστασίας. Διότι η προστασία αφενός θα πρέπει να δει τι οργανισμοί υπάρχουν ήδη, παραδείγματο χάρη επιτροπές για ανηλίκους, ε, αλλά που θα, για τα μέσα ενημέρωσης που θα επικεντρώνονται φυσικά και στα ψηφιακά μέσα και από εκεί και πέρα θέματα παρόχων, υπηρεσιών και εκπαιδευτικών οργανισμών. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι αυτό που προκύπτει από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία μορφία μεταξύ των κρατών μελών. Ε, χωρίς όμως λοιπόν εμείς να περιορίσουμε την επικουρικότητα, να δούμε το θέμα από κοινού όσο γίνεται και να προσπαθήσουμε και σε κοινοτικό επίπεδο να έχουμε μία προσέγγιση που θα είναι πιο ε, οργανωμένη. Δεύτερο ζήτημα Πρώτο θέμα λοιπόν η διακυβέρνηση με, από όλε τι πτυχέ. Δεύτερον, πώ μπορούμε να προάγουμε το δικαίωμα στην πρόσβαση και στην παιδεία για τα μέσα ενημέρωση. Το να είμαστε λοιπόν ε, να μην είμαστε ψηφιακά αναλφάβητοι, διότι πλέον αυτό είναι θέμα βασικής παιδείας και όπως πλευρέπει η ψηφιακή ατζέντα να περιλάβουμε όλες αυτές τις ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις ε, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να χρωματοδοτούνται και αυτά τα προγράμματα μαζί με τα υπόλοιπα. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο και προκύπτει από όλες τις οργανώσεις με τις οποίες ήρθα σε επαφή, διότι είχαν αρκετές διαβουλεύσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με υπευθύνου για το πρόγραμμα Safer Internet που ε, είναι όλοι ενταγμένοι σε ένα ευρύτερο δίκτυο που λέγεται Naxos, το European Net που περιλαμβάνει περιλαμβάνει αρκετέ ευρωπαϊκέ χώρε, πολλέ λοιπόν μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά και παραγωγού ηλεκτρονικών παιχνιδιών, διαδικτυακών παιχνιδιών και ε, παρόχου ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύ μεγάλο ε, αμάλγαμα οργανώσεων και αυτό το οποίο προέκυψε σαφώ ε, και το ζητά και ο κόσμο των επιχειρήσεων και των ε, ε θεσμικών οργάνων όμω, είναι να υπάρχουν κάποιε εκπαιδευτικέ συμμαχίε πολύ πιο στεναρές ε, οργανώσεις ε, ε, εκπαιδευτικών αλλά και γονέων και κυδεμόνων. Το θέμα των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικό, αλλά φυσικά και οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα ανηλίκων αλλά και με επιχειρήσεις. Μία πολύ σημαντική καινοτομία την οποία επισημαίνω διότι θεωρώ ότι θα πρέπει να την προωθήσουμε και να ζητήσουμε την εφαρμογή της είναι η πρόσφατη συμφωνία που έκανε η Επίτροπος Κρόους ε, τον Ιανουάριο του 2012, πριν από ένα μήνα δηλαδή, με τη λεγόμενη CO Coalition. Πρόκειται για μια συμφωνία την οποία προσυπογράφουν προς το παρόν 25 επιχειρήσεις ε, στο ψηφιακό κόσμο. Αναφέρομαι στους παρόχους υπηρεσιών, που είναι πάροχοι είτε ηλεκτρονικών υπηρεσιών είτε πάροχοι διαδικτύου και υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ των δύο και υπάρχει αυτή η συμφωνία που είναι μια πολύ καλή άγουσα και η έκθεσή μου θα ήθελε να προωθηθεί και από πλευρά κρατών μελών και να εφαρμοστεί στη συνέχεια η οποία προβλέπει πέντε στόχους πάρα πολύ σημαντικούς και που ενδιαφέρουν και όλες οι οργανώσεις που άκουσα. Ε, πρώτον, notice and take down, δηλαδή εάν ε, υπάρχει παράνομο ή επιζήμιο περιεχόμενο, μόλις κοινοποιείται θα πρέπει να κατεβαίνει στο σελίδα. Υπάρχει και μία σχέση με την οδηγία για την παιδική πορνογραφία και αναφέρομαι μόνο στο παράνομο περιεχόμενο. Πράιβαση από εκεί και πέρα, ιδιωτική ζωή. Ε, μιλώντας με τον Ευρωπαίο ε, υπεύθυνο για θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, θα υπάρχει και εμπλοκή του Ευρωπαίου υπευθύνου ε, και η Επίτροπος Ρέτινγκ έχει αναφέρει ότι θα υπάρχει μια οδηγία πολύ ενδιαφέρουσα για το θέμα ε, ε, της ιδιωτικής ζωής ε, και θα πρέπει να δούμε τι σχέση υπάρχει με αυτό. Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος από πλευράς γονέων. Αυτές που σας αναφέρω είναι οι πέντε αρχές. Ε, τα στάνταρ από εκεί και πέρα για τα τέτοια κατάχρηση για να δούμε κατά πόσον υπάρχουν καταχρήσεις με κάποιο πιο ομογενή τρόπο και από εκεί και πέρα συστήματα αναγνώρισης. Είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το τελευταίο ζήτημα διότι υπάρχουν νέες μορφές κατάχρησης ε, και ε, κακοποίησης ανηλίκων που χρησιμοποιούν πιστοτικές κάρτες οι οποίε κατά πάσα πιθανότητα είναι των γονέων, αλλά τα παιδιά ε, έχουν κατοχή των καρτών αυτών και ε, χρησιμοποιούν τον αριθμό για να παίξουν ηλεκτρονικά παιχνίδια από εκεί και πέρα στο διαδίκτυο, που κάποιε φορέ είναι και παράνομα ή επιζήμια για την υγεία του και γενικώ ε, προβληματικά. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και τα θέματα ηλικίας, κατάλληλη ηλικία για την πρόσβαση. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, για παράδειγμα, υπάρχει απαγόρευση, δεν μπορούν να πολλούνται παράνομα ηλεκτρονικά παιχνίδια και ε, ε, ο έμπορος έχει κυρώσει, ενώ για τα διαδικτυακά παιχνίδια το μόνο φίλτρο που υπάρχει είναι να υπάρχει μια πιστοτική κάρτα η οποία θα πρέπει να είναι ε, ε, ιδιοκτησία ενός ενήλικα. Ε, υπάρχουν λοιπόν κάποια θέματα διαδικτύου τα οποία θα πρέπει να ελέγξουμε και μπορεί να υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι και να αποτελούν ε, πρόβλημα για την ιδιωτική ζωή των παιδιών. Προσπάθησα λοιπόν να κάνω μία διάκριση μεταξύ των θεμάτων που σχετίζονται με πτυχές που είναι παράνομες ή πτυχές οι οποίες είναι επιζήμιες ή ακατάλληλες. Είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο παράνομο, διότι δεν αναφερθήκαμε καθόλου στο θέμα της παιδικής ε, πορνογραφίας, διότι ρυθμίζεται από άλλη οδηγία, προσπάθησα να επισέλθω σε μία άλλη φαιά ε, περιοχή. Ε, για παράδειγμα, πορνεία στο διαδίκτυο, ε, μορφές ε, ε, παραπλάνησης, grooming, όλα αυτά είναι επιζήμια και τα οποία μπορεί να έχουν και πολύ μεγάλους κινδύνους και για την σωματική και φυσική ψυχική ακεραιότητα των παιδιών και όλα αυτά τα θέματα είναι πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε με ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά θα πρέπει να τους δώσουμε τη δέουσα προσοχή. Αυτό λοιπόν ε, είναι για τα θέματα της προστασίας. Όσον αφορά τώρα την προαγωγή της ε, υπηκότητας, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και θα ήθελα επ' αυτού να κάνω κάποιες πολύ συγκεκριμένε αναφορές σε προγράμματα τα οποία είναι ήδη εν εξελίξη ε, και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία η ηλεκτρονική δημοκρατία, η ηλεκτρονική συμμετοχή και όχι μόνο το να είναι κάποιος ψηφιακά γνώστης κάποιων πραγμάτων, ε, και μέσω αυτών των προγραμμάτων τα παιδιά μπορούν να δουν πώς λειτουργεί η δημοκρατία, να μπορούν ε, για παράδειγμα να ε, ορίσουν έναν προϋπολογισμό ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν είδη παιχνιδιού όλα αυτά. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Ε, υπάρχει ένα πρόγραμμα, πάνω από 30 χώρες συμμετέχουν σε αυτό το ε, πρόγραμμα δικτύο Schoolnet. Υπάρχουν λοιπόν και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 30 ε, ευρωπαϊκές χώρες, που δημιουργεί έναν ψηφιακό κοινό ε, σχολικό χώρο. Και εδώ κάνω μια πρόταση από αυτού, διότι αν δεν κάνω λάθος από αυτά που άκουσα από τις οργανώσεις και από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι ήδη όριμη η κατάσταση και μπορούμε να προωθήσουμε και τη δημιουργία κάποιου κοινωνικού φόρουμ, τα οποία θα έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και μπορούν να δημιουργήσουν και αδελφοποιήσεις όπως γίνεται γίνεται ήδη μεταξύ σχολείων σε έναν ψηφιακό χώρο πλέον. Ε, στην ουσία, και αυτή είναι και η πρότασή μου, είναι να δημιουργήσουμε εκ νέου το πλαίσιο που δημιουργήθηκε και να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα νέα μέσα ενημέρωσης και ταυτόχρονα να έχουμε προστασία των ανήλικων χρησιμοποιώντας την νομοθεσία που έχει αλλάξει πολύ το τελευταίο διάστημα, αλλά ταυτόχρονα να διερευνήσουμε μέσω τη προσέγγιση αυτή, τη διακυβέρνηση, τη παιδεία, τη ενεργού συμμετοχή, τη υπηκότητα και της νέε μορφές προστασίας, ε, αυτές τις περιοχές οι οποίες είναι πολύ θετικέ και πολλά υποσχόμενε, αλλά και τι φαίε ζώνε, οι οποίες ε, ε, δεν καθορίζονται σαφώ, διότι υπάρχει παιδική πορνογραφία η οποία είναι σαφώ ορισμένη, αλλά υπάρχουν και οι άλλε μορφές, οι οποίες μπορεί να είναι άλλε μορφές κακοποίησης ή κατάχρηση. Ε, από εκεί και πέρα ε, οι χώρες μέλη, κάποιες πιο προηγμένες, κάποιες λιγότερο προηγμένες, ε, που έχουν συγκεκριμένες μορφές ε, ε αυτορύθμισης, συμφωνιών ή συρρύθμισης, ε, μπορούμε μέσω αυτών των μορφών να πάμε σε πιο στεναρές μορφές παρέμβασης. Αυτό προείπησε και από άλλες συζητήσεις. Στη χώρα μου και σε όλες χώρες υπάρχει και η δυνατότητα να μπλοκάρονται κάποιες ιστοσελίδες. Σε κάποιες άλλες χώρες δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει δυνατότητα αφαίρεσης περιεχομένου πολύ γρήγορα. Υπάρχει λοιπόν και το θέμα Τη της των παρόχων των υπηρεσιών που είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει σε κρεμότητα. Θα κάνω κάποιες προτάσεις από αυτό και θα δω κατά πόσο θα τις ημερίζεστε κι εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, για τα σχόλια σας, κύριε Κώστα. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. είναι τόσες πολλές δυνατότητες του ίντερνετ που φέρνουν και πολλούς κινδύνους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 41% των παιδιών μεταξύ 12 και 15 ετών έχουν smartphones και τα χρησιμοποιούν και καθημερινά. Τεράστιο ποσοστό. Και 48% από αυτά τα παιδιά που, τα χρησιμοποιούν τα smartphones ε, δεν είναι πολύ ευχαριστημένα με το περιεχόμενο το οποίο βρίσκουν στο ίντερνετ. Όμως ε, ασφαλώς ε, έχουμε πολλές ε, ευκαιρίες αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τους κινδύνους για τους ανήλικους. Το ακατάλληλο περιεχόμενο, το grooming, την παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση κλπ. Και η κοινωνική δικτύωση επίσης πολλές φορές χρησιμοποιει σε πολλούς ε, νέους ε, για να ε, διαχειριστούν τις σχέσεις τους με άλλους ανθρώπους, πράγμα που δημιουργεί πολλά προβλήματα συχνά. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε και περιπτώσεις αυτοκτονίας για γεγονότα που συνέβησαν διαδικτυακά. Ασφαλώς το κλειδί είναι οι δάσκαλοι και οι γονείς να ευαισθητοποιούν τα παιδιά τους και οι γνώσεις, περισσότερες γνώσεις για το διαδίκτυο και τις τεχνολογίες επίσης θα βοηθήσουν. Ασφαλώς και οι πάροχοι ε, θα έχουν να παίξουν το ρόλο τους και τα ίδια τα ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχουν κάποια εργαλεία, θα πρέπει να τα γνωρίζουμε. Για παράδειγμα το μπλοκάρισμα διευθύνσεων και ε, σελίδων που έχουν περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας, καθώς επίσης και εργαλεία για να αντιμετωπιστούν τα δίκτυα παιδικής ε, ε, ε, πορνείας. Χρειάζονται όμως περισσότερες δράσεις και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Χρειάζεται να ε, χρησιμοποιήσουμε ένα μείγμα ε, αυτορύθμισης και νομοθεσίας. Και θα πρέπει να είναι ένα μείγμα το οποίο θα προσαρμόζεται στην πραγματικότητα. Πάντως σίγουρα θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές μας λύσεις, αλλά θα πρέπει να κάνουμε κάτι έτσι ώστε τα παιδιά ε, να εποφελούνται πραγματικά του χρόνου που περνούν στο διαδίκτυο χωρίς ε, να υφίστανται τους κινδύνους του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Πέτρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ και την Σίλβια για την παρουσίαση του θέματος αυτού η προστασία των νέων στο διαδίκτυο είναι από τα πιο δύσκολα προβλήματα τα οποία θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε και όλοι αυτοί που έρχονται από τη Γερμανία γνωρίζουν ακριβώς τη συζήτηση που έχει λάβει η χώρα τον προηγούμενο και τον πιο προηγούμενο χρόνο στη Γερμανία και οι προσπάθειες αυτές να καταλήξουμε σε μια συμφωνία απέτυχαν γιατί είναι πολλές οι διακλαδώσεις και οι επιπτώσεις στα θέματα αυτά, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεγονός ότι η γνώση των μέσων των διαδικτυακών είναι το κλειδί για τη λύση. Θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ βλαβερού περιεχομένου και παρανόμου περιεχομένου. Το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να σβήνεται αμέσως από το διαδίκτυο. Για το βλαβερό περιεχόμενο όμως μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συζήτηση πολύ γρήγορα η οποία και σε κάθε χώρα μέλος έχει διαφορετικό χαρακτήρα γιατί όλα αυτά εξαρτώνται από την πολιτιστική παράδοση κάθε χώρας. Βλέπουμε ότι το σύστημα της ε, αυτορύθμισης είναι κάτι το οποίο θεωρούν ορισμένοι ότι μπορεί να καλύψει αυτά τα θέματα. Αλλά παραδείγματο χάρη τα όρια ηλικία διαφέρουν από μια χώρα στην άλλη. Μπορεί να είναι 14 χρόνια σε μια χώρα, 16 στα άλλα. Υπάρχουν ήδη μεγάλε πολιτιστικέ διαφορέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα θέματα αυτά και σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του τι είναι βλαβερό περιεχόμενο και το τι δεν είναι. Επομένω θα πρέπει να προσέξουμε ότι υπάρχει αυτή η πολιτιστική πολυμορφία η οποία είναι δικαιολογημένη λόγω της παράδοσης και δεν θέλουμε να τα ισοπεδώσουμε όλα, πρέπει να βρούμε μια λογική λύση. Και όταν μιλάμε για την ικανότητα αντιμετώπισης των ψηφιακών μέσων, δεν πρέπει να μιλήσουμε μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς και την ευθύνη που έχουν οι γονείς σε σχέση με τα θέματα αυτά. Γιατί ιδιαίτερα για τους ε, ενήλικες να θέσουμε την έμβαση και φυσικά θα πρέπει να έχουμε μια όλος ιδιαίτερη έμφαση στα μέσα κοινωνικής διαδικτύωσης, τίθενται επίση τα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτά ανήκουν σε ένα άλλο τομέα. Πάντα όμως θα πρέπει να έχουμε αυτό το στοιχείο το οποίο έχει να κάνει με την παιδική πορνογραφία. Γιατί δεν θέλουμε να καλύψουμε την παιδική πορνογραφία από την ελεύθερη έκφραση στο διαδίκτυο και να εμποδίσουμε τον έλεγχο των διαδικτυακών ροών. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε ένα πολύ συγκεκριμένο επίπεδο και ελπίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή καλή λύση η οποία εξυπηρετεί την προστασία των παιδιών, κάνει <clears throat> πάντα δυνατό το να μπορούν οι νέοι και τα παιδιά να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, αλλά και αντιμετωπίζει τις ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν για την ελευθερία έκφραση στο διαδίκτυο και την ελευθερία πρόσβαση στην πληροφορία, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν πρέπει να περάσει στο περιθώριο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένας ελεύθερος χώρος επικοινωνίας και αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όταν μιλάμε για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να βρούμε το, την κατάλληλη ισορροπία. Ευχαριστώ Πέτρα. Η Μαρία έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα είμαι σύντομη γιατί έχουν ελεχθεί περί τα περισσότερα από αυτά που ήθελα να πω. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την συγγήτρια. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Και υπάρχουν, αν θέλετε, και μερικές προφανείς λύσεις <clears throat> που είναι καταρχήν να υπάρχουν για τους νέους ορισμένα φίλτρα από, το, ε, από εξ αρχής, χωρίς δηλαδή να υπάρχει καμιά παρέμβαση για να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θέλω να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι το ε, ανεπιθύμητο περιεχόμενο δεν είναι το ίδιο πράγμα με το παράνομο ή το βλαβερό περιεχόμενο. Μπορεί ο καθένας να ορίσει το ανεπιθύμητο περιεχόμενο με, τους, με το δικό του τρόπο. Μπορεί κάποιος για λόγους συμφερόντων να μην κάνει μια αμερόληπτη αξιολόγηση του τι είναι ανεπιθύμητο ή όχι. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι ε, ικανοί οι Ευρωπαίοι πολίτες, μικροί και μεγάλοι, σε θέση να κάνουν σωστά πληροφορημένες και εμπεριστατωμένες αποφάσεις. Έχουν λεχθεί πάρα πολλά για την αυτορύθμιση του τομέα αυτού του διαδικτυακού. Εγώ δεν υποστηρίζω την υπερβολική ρύθμιση, δεν υποστηρίζω το να δημιουργήσουμε νέα στρώματα, νέες στρώσεις γραφειοκρατίας ή να έχουμε το μεγάλο αδερφό της κυβέρνησης να παρεμβάνει στην προσωπική ζωή των ανθρώπων. Αλλά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα τα θέματα αυτά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για το ποιος θα αστυνομεύει το διαδίκτυο γιατί ο τρόπος με τον οποίο ε, εκπονούμε κανόνες για όλα αυτά δίνει και ένα μήνυμα στην επόμενη γενιά. Και φτάνουμε σε βασικές έννοιες μιας ανοιχτής δημοκρατίας. Είναι ο δικαστής ο οποίος κρίνει αν μια πληροφορία είναι παράνομη ή όχι ή είναι μια εταιρεία. Και αν είναι μια εταιρεία ποιες είναι οι παράπλευρες ζημίες που μπορούν να προκύψουν. Κάποιος ο οποίος είναι ακτιβιστής ως εταιρεία δεν θα πιέσει υπερβολικά στο να αφαιρείται κάποιο περιεχόμενο. Ποιος θα είναι υπεύθυνο για αυτή την απόφαση και ποιος μπορεί να υποφεληθεί από τέτοιου είδου αποφάσεις. Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε και τον διαχωρισμό των εξουσιών και την δημοκρατική εποπτεία για να υπάρχει σωστή εποπτεία της λήψης αποφάσεων. Είδαμε ότι υπάρχει μια ολιστερή κατοφέρεια για τα θέματα αυτά. Το κόμμα μου έθεσε ένα ερώτημα στην Κομισιόν πέρσι όταν ετέθη το θέμα για το μπλοκάρισμα ορισμένων ιστοσελίδων στο ίντερνετ για να, να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν είναι για ένα θέμα μπλοκαρίσματος της παιδικής πορνογραφίας. Αυτό συμφωνούμε όλοι ότι αυτό πρέπει να γίνεται. Αλλά μήπως το μέτρο αυτό του μπλοκαρίσματος των ιστοσελίδων μπορεί να προχωρήσει σε άλλες περιοχές από το παράνομο περιεχόμενο να μπούμε στο ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Μήπως η μουσική παραγωγή, παραγωγή χάρη, θα θελήσουν να κατέβουν ορισμένες, ε, ορισμένοι στο χώρο κτλ. Η Κομισιόν μας είπε όχι μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένας λόγος για κάτι τέτοιο να ανησυχείτε, αλλά πρόσφατα γεγονότα μας κατέδειξαν ότι οι ανησυχίες αυτές είναι ανησυχίες που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη σοβαρά. Είδαμε να κατεβαίνουν οι στόχοροι χωρίς παρέμβαση δικαστικής εξουσίας επί τη βάση μονάχα των Αμερικανικών ε, δικαστικών διαδικασιών που μπορούν να έχουν επίπτωση σε όλο τον κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση έχει πολλές σημαντικές πτυχές και ελπίζω, εύχομαι κάθε επιτυχία στην εισηγήτρια, ελπίζω να βρει τη σωστή ισορροπία. Θέλω να υπογραμμίσω όμως ότι ακόμα και αν το παράνομο ή το ανεπιθύμητο περιεχόμενο δεν είναι πια ε, ορατό στο ίντερνετ, αυτό σημαίνει, δεν, δεν σημαίνει ότι έχει εξαφανιστεί, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα και δεν σημαίνει ότι η λύση που έχουμε βρει είναι βιώσιμη. Επομένως θα πρέπει να βλέπουμε πάντα την πλήρη εικόνα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σανίτσι. Κυρία Σανίτσι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Συγχαίρω την κυρία Κώστα για την παρουσίαση, ιδίω για τα θέματα προστασία ε, των ανηλίκων στον ψηφιακό κόσμο. Και συμφωνώ απολύτω μαζί τη σε όλα. Πολύ καλή δουλειά, πράγματι. Τα τελευταία χρόνια ο ψηφιακό κόσμο ε, είναι πιο σημαντικό ακόμα και ε, από την τηλεόραση και η συμμετοχή στο διαδίκτυο των ανηλίκων είναι καθημερινά στην ε, ε, ζωή τους και μπορεί να επηρεάσει και τους ίδιους αλλά και τις συμπεριφορές τους. Ξέρουμε ότι δεν θα επικεντρωθούμε στην παιδική προγνωγραφία στο διαδίκτυο διότι επί του ζητήματος έγιναν συζητήσεις και υπήρξε και σχετική έκθεση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Αλλά όπως εξήγησε πάρα πολύ καλά η κυρία Κώστα υπάρχουν θέματα δικαιώματο πρόσβασης και δικαιώματος στην προστασία τα οποία είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να διασφαλίσουν ότι οι νέοι θα έχουν ε, πρόσβαση σε ασφαλείς ιστοτόπους και θα προστατεύονται από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να προσπαθήσουμε να βρούμε όλες τις πολιτικές που θα μπορέσουν να νικήσουν την εξάρτηση και την απώλεια της, αίσθηση της αίσθησης της πραγματικότητας και της μοναξιάς που ε, προκύπτουν από την πάρα πολύ μεγάλη παραμονή στο διαδίκτυο. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην κυρία Κώστα. Ε, έχει την πλήρη υποστήριξή μου και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τη βοηθήσω. Ευχαριστώ. Mr. Boris. Ο κύριος Μπόρις. Ευχαριστώ. Να ε, ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση, η οποία πραγματικά είναι κέρια δεδομένων των δραστηριοτήτων μας ε, για την ελευθερία στο ίντερνετ. Πρέπει ταυτόχρονα να προστατεύσουμε και την ε, νέα γενιά που πλέον απομακρύνεται κατά σε κάποιο βαθμό από τις ε, πραγματικές διαπροσωπικές σχέσεις προς όφελος των σχέσεων μέσω του κυβερνοχώρου. σε, στον δημόσιο διάλογο και στην ε, δημόσια εκπαίδευση θα μπορούσαμε ε, να λάβουμε υπόψη αυτή τη διάσταση έτσι ώστε να προετοιμάζουμε τα παιδιά για τα νέα μέσα ε, επικοινωνίας και το ίντερνετ. Οι δάσκαλοι καταρχήν που είναι μοντέλα για τα παιδιά, μοντέλα προς αντιγραφή για τα παιδιά, <laughs> δεν ξέρουν πολύ συχνά ε, να χειρίζονται τις τεχνολογίες αυτές και δεν ξέρουν τι σημαίνει στο ίντερνετ. Συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενημερωθούν οι ίδιοι δάσκαλοι, οι ίδιοι καθηγητές ε, και όχι μόνο τα παιδιά. Το άλλο που πρέπει να διοργανώσουμε είναι ε, εκστρατείες γενικότερα κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Η οικογένεια, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ σημαντική για τα παιδιά, η επαφή των παιδιών με τους γονείς. Και εκεί πάλι έχουμε ένα τεράστιο χάσμα γενεών, γιατί οι γονείς πολλές φορές ε, δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις τεχνολογικές εξέλιξεις. Οπότε δεν καταλαβαίνουν καν τι κάνουν τα παιδιά στο ίντερνετ και δεν καταλαβαίνουν σε τι περιεχόμενο έχουν τα παιδιά τους πρόσβαση. Οπότε θα πρέπει οι γονείς, τους να, οι γονείς να μιλάνε με τα παιδιά τους και να τα ενημερώνουν, να τα προειδοποιούν για τους κινδύνους. Τα περισσότερα εθνικά στήματα εκπαίδευσης ε, δεν λαμβάνουν υπόψη αυτόν τον παράγοντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια γιατί νομίζω ότι την περιμένει δύσκολο έργο και πρέπει να πω ότι μου πήρε τα λόγια από το στόμα ο κύριος Μπόρις, διότι συμφωνώ πολύ με τα όσα είπε υπό την έννοια ότι θεωρώ ότι υπάρχουν δύο ε, μορφές προβλημάτων. Καταρχάς ε, το νομοθετικό πλαίσιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τα κατάλληλα νομικά μέσα για την προστασία των ενηλίκων, διότι ο τεχνολογικός κόσμος εξελίσσεται τόσο γρήγορα που κάθε χρόνο έχουμε νέες τεχνολογίες και θα ήταν μάλλον δύσκολο να μπορέσουμε να προστατεύσουμε από νομική σκοπιά στους ανηλίκους σε ένα τέτοιο ζήτημα. Και μάλιστα διαπιστώνουμε ότι κάθε χώρα έχει τελείως διαφορετική νομοθεσία η οποία ε, δεν είναι καν όμοια μεταξύ της ούτε εντό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και τα θέματα της ευαισθητοποίησης στο σχολικό περιβάλλον αλλά και δυστυχώς και στην οικογένεια. Και λέω δυστυχώς διότι το χάσμα των γενεών επιτείνει το πρόβλημα. Οι γονείς πολλές φορές δυσκολεύονται να καταλάβουν τι είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι νέες τεχνολογίες, το διαδίκτυο και τι κινδύνους ε, έχει και πού μπορεί να φτάσει. Επομένως θα πρέπει να γίνει μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και εντό των οικογενειών για τους γονείς για να μάθουν ποιοι είναι οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους ορισμένες φορές στο διαδίκτυο ε, διότι πολλέ φορές απουσιάζουν και οι γνώσεις για να κατανοήσουμε τι κίνδυνοι ελοχεύουν ε, σε αυτές τις νέες μορφές τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων. thank you, Mr. Fontana. Now I would like to... Ευχαριστώ κύριε Φοντάνα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν αν θα ήθελε να λάβει το λόγο ή εκπρόσωπος της Κομισιόν κυρίως. Σας ευχαριστώ. Χαιρετίζουμε την απόφαση του Κοινοβουλίου να προχωρήσει σε μια έκθεση για τα θέματα αυτά. Η συζήτηση εξήρε ορισμένα σημεία τα οποία θα ήθελα και εγώ να τονίσω και να διευκρινίσω στο βαθμό του δυνατού. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει από τα ερευνητικά στοιχεία ότι υπήρξε μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που τα παιδιά και οι νέοι χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες. Βλέπουμε ότι τα παιδιά περνάνε στο διαδίκτυο σε όλο και μικρότερη ηλικία, ήδη από τα 7 σε ορισμένε χώρες, αλλού ακόμα νωρίτερα. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη έκθεση στο διαδίκτυο που οδηγεί και στην ανάδυση νέων κινδύνων, όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, κινδύνοι που έχουν να κάνουν με βλαβερό ε, περιεχόμενο, με grooming, με απώλεια της ιδιωτικότητας κτλ. Βέβαια δεν υπάρχει πάντα το κατάλληλο περιεχόμενο υψηλής ποιότητας για τα παιδιά στο διαδίκτυο και όπως είπανε πολλοί ομιλητές εξακολουθεί σε πολλές περιπτώσεις να υπάρχει υλικό παιδικό πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Όπως είπε και η συγγήτρια σωστά, η Κομισιόν έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα για το ασφαλές ε, διαδίκτυο, το οποίο θα λειτουργεί ακόμα μέχρι το 2013 και έχουμε σημαντικά επιτέγματα στο πρόγραμμα αυτό. Υπήρξε ένα δίκτυο ασφαλών κέντρων ίντερνετ σε όλα τα κράτη-μέλη. Περιλαμβάνουν και μια γραμμή επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης και έχουν πολλές από τις ε, δυνατότητες που ανέφεραν και άλλοι ομιλητές να υπάρχουν ε, μαθήματα, εκπαίδευση, συνειδητοποίηση των παιδιών και των γονέων. Το 2010 έγινε μια μεγάλη έρευνα για τα παιδιά και τους γονείς σε 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε μια πολύ καλή δυνατότητα ενόρασης στις νέες εξελίξεις στα θέματα αυτά. Αυτό που μας δείχνει αυτή η έρευνα είναι ότι πρέπει να βρούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τη ρευστότητα του τομέα αυτού και τις συνεχείς αλλαγές. Είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουμε πάντα ενήμεροι σε νομοθετικό επίπεδο. Προς το παρόν λοιπόν η Κομισιόν προτείνει με το πρόγραμμα του ασφαλούς ίντερνετ να να συνεχίσουμε και τη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος και του προγράμματος Connect Europe Προτείνει λοιπόν η Κομισιόν μια σειρά αποδράσεις που βοηθάνε την ασφάλεια στο ίντερνετ για τα παιδιά και η Κομισιόν προτείνει να επενδύσουμε σε κοινού και διαλειτουργικούς πόρους να υποστηρίξουμε το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Ασφαλών Κέντρων Ιντερνετ σε όλη την Ευρώπη και να διαμοιραστούμε τους πόρους για να υπάρχει καταγραφή αυτών οι οποίοι παραβιάζουν την νομοθεσία περί πορνογραφίας κτλ. Επίσης θα πρέπει να αυξήσουμε την κλίμακα αυτών των δραστηριοτήτων και μας ενδιαφέρει να υπάρξει και η οικειοποίηση αυτών των ε, πληροφοριών, πώς μπορούν να κάνουν ευφύς, να παίρνουν ευφύς αποφάσεις οι γονείς και τα παιδιά όταν βρισκόνται στο διαδίκτυο. Θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε το περιεχόμενο ποιότητα στο διαδίκτυο για θέματα όπως είναι η ιδιωτικότητα. Η Κομισιόν έχει υποβάλει μια πρόταση για την προστασία των δεδομένων μέσα στον κανονισμό αυτό και συγχρόνως, όπως είπαν και ορισμένοι προηγούμενοι ομιλητές, η Κομισιόν υποστηρίζει την αυτορύθμιση του τομέα αυτού στο διαδικτύου. Η συγγήτρια ήδη αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία την, το συνασπισμό αυτών που ξεκίνησε η Επίτροπος Κρούζ το 2011. Υπάρχουν 30 επιχειρήσεις που συμμετέχουν και καλύπτουν ε, τις εταιρείες κοινικής τηλεφωνίας, τους κατασκευαστές κινητών συσκευών, τους παρόχους υπηρεσίες κτλ. Αλλά είναι και μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, διοκτικές και αστυνομικέ αρχές ε, κτλ. ώστε να συζητήσουν από κοινού όλα αυτά τα θέματα που αναφέρει η, η συγγήτρια, να υπάρχουν φίλτρα κατάλληλα με την ηλικία, να υπάρχει μεγαλύτερη χρήση γονικών ελέγχων και επίσης και καταστροφή ιστοσελίδων που έχουν καταχρηστικά για τα παιδιά περιεχόμενα. Προσπαθούμε λοιπόν να προχωρήσουμε προς την εφαρμογή όλων αυτών των δράσεων και ελπίζουμε ότι θα έχουμε περισσότερα στοιχεία το καλοκαίρι. Είμαστε πάντα σε επαφή με την κυρία Κώστα και περιμένουμε να ακούσουμε και την τελική θέση του Κοινοβουλίου. Κυρία Κώστα, θέλετε να λάβετε το λόγο. Δύο λόγια μόνο. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, φυσικά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, διότι κατανοώ ότι το ζήτημα είναι ευαίσθητο, αλλά νομίζω ότι μας αφορά λίγο όλους. Ε, υπάρχει ένα αίσθημα ευθύνη προς ένα ζήτημα το οποίο ε, εξετάζει για πρώτη φορά ε, στην ιστορία της γνώσης τόσες πολλές δυνατότητες ταυτόχρονα και τόσους πολλούς κινδύνους. Αυτή είναι η δυσκολία αυτού του θέματος. Δεν μου διαφεύγει, το λέω και για τους αδέλφους που τα ανέφεραν, ο κύριος Μπόρης, ο κύριος Φοντάνα, η κυρία Σάκη, η κυρία Τζανίκη. Είναι σαφές ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται μπροστά μας. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ε, το είπε και η κυρία Καμερέβερ. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βρούμε ένα σημείο ισορροπίας και το σημείο ισορροπίας δεν είναι μόνο ένα σημείο ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας της ενημέρωσης, της έκφρασης ε, και των συμπεριφορών αλλά και της κατάλληλης προστασίας. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αυτά τα δικαιώματα είναι εγγενή δικαιώματα και της Χάρτας ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ε, που είναι πλέον εγγεγραμμένη ε, στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Και μάλιστα στη Συνθήκη της Λισαβόνας η προστασία των ανηλίκων είναι αναπόσπαστο στοιχείο του συντάγματος. Και το αναφέρει αυτό ρητά η συνθήκη της Λισαβόνας. θα πρέπει λοιπόν πέρα από το δικαίωμα της έκφρασης προς τους ανηλίκους και το δικαίωμα της συμμετοχής, να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανηλίκους αφενός να προστατεύουμε την ανθρώπινη τους αξιοπρέπεια αλλά και τη δυνατότητα να αναπτυχθούν κατάλληλα σε ψυχοσωματικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία που αφορούν και τους ανηλίκους αλλά ε, και τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να έχουμε κατά νου. Γνωρίζω πολύ καλά τι συζήτηση έγινε για την παιδική πορνογραφία, όπου όλα τα θέματα τα οποία ε, αφορούσαν και τις πολυπολιτισμικές ε, ε, διαφορές ε, και τις διάφορες ηλικιακές ομάδες και ούτε καθεξής. Αλλά εδώ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νομοθεσία, έχουμε μία έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ πρέπει να έχουμε κατά νου ότι πάντα υπάρχει κατάχρηση όταν δεν υπάρχουν οι υποκειμενικές ή αντικειμενικές συνθήκες οι οποίες επιτρέπουν σε ένα ανήλικο παιδί να εκφραστεί πλήρως. Αυτή είναι η δυσκολία όταν μιλάμε για ανηλίκους. Πέραν αυτού όμως, ε, θα προσπαθήσω να λάβω πολύ σοβαρά υπόψη ε, τα όσα μας είπατε και φυσικά και τους ε, διάφορους όρους που πρέπει να θέσουμε ώστε να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε όλα τα ζητήματα μεταξύ των. Θα πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί ε, ε όντας ψηφιακά ενήμοροι και ορισμένε φορές γνωρίζουν πολύ περισσότερο και από τους γονείς τους ε, είναι πάντα αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Ε, υπάρχουν όμως κάποιες φορές όπου μπορούμε να έχουμε και εμπορική εκμετάλλευση του ατόμου του ανηλίκου. Αναφερόμαστε όμως και σε μια απόλυτη καινοτομία των τελευταίων χρόνων που είναι η σύγκληση μεταξύ των συστημάτων. Μεταξύ ενός κινητού τηλεφώνου μέσω ενός iPhone ο ανήλικος πλέον μπορεί να έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες έκφρασης και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μπορούμε να ρυθμίσουμε και όλα αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα λοιπόν να λάβουμε υπόψη και να υπάρχει και αυτό στην έκθεση ε, ότι υπάρχουν δύο κώδικες εντολογίας ε, πολύ σημαντικοί. Ένας ε, για την κινητή τηλεφωνία και ένας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία και θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχες συμφωνίες κατά την άποψή μου και σε επίπεδο κρατών μελών. Επίσης, ο χώρος κοινωνικοποίησης, όπως έλεγε η κυρία Τζανίκη, είναι πλέον το διαδίκτυο. Επομένως υπάρχει και πρόβλημα ενημέρωσης μπορεί να υπάρχουν κάποιε προειδοποίησει και προ του γονεί, αλλά και προ τα ίδια τα παιδιά. Υπάρχουν κάποιε ιστοσελίδε, γνωρίζω στην Ιταλία με πολύ ενδιαφέρουσα, ε, πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα που γίνεται από εφήβου. οι οποίοι εφήβοι ενημερώνουν του ίδιου του συνομιλίκου του και του λένε για παράδειγμα προσέξτε το τάδε ή ε, προσπαθούν να του βοηθήσουν να κατανοήσουν πώ ακριβώ να κινηθούν σε αυτέ τι ιστοσελίδε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το σχολείο τώρα. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πράγματι, μπορεί κάποιο να ξεκινάει και από 7 χρονών, αλλά υπάρχουν παιδάκια 4 χρονών που έχουν ψηφιακέ δεξιότητε ενώ δεν ξέρουν καν να γράφουν ακόμα. Επομένω, το σχολείο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια νέα ομάδα στόχων παιδιών που έχουν μια δεξιότητα ε, σαν να ξέρουν να διαβάζουν. Ξέρουν ήδη πώ είναι οι διάφορε ιστοσελίδε και λένε στου γονεί του τι πρέπει να κάνουν για να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο ενώ ακόμα δεν ξέρουν να γράφουν το όνομά του. Πρόκειται λοιπόν για νέε δεξιότητε, τι οποίε όλοι καλούμαστε να απαντήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ήδη από το σχολείο να υπάρχει πολύ πιο συγκεκριμένη δράση και πρέπει να ζητάμε όπω γίνεται και από την ψηφιακή ατζέντα ε, αλλά να το κάνουμε και στην έκθεση να ζητήσουμε λοιπόν να συμπεριληφθεί το θέμα θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και ε, την προσφορά ποιότητας και στα διδακτικά μέσα στα πλαίσια του σχολείου ε, και να είναι αυτά πλέον καθήκον και όχι μόνο μια δυνατότητα επιλογής στα σχολικά προγράμματα. Και μέσω και των διαρθρωτικών ταμείων να υποστηρίξουμε αυτή την επέκταση αυτών των αρμοδιοτήτων και να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πλέον αυτά τα μέσα επικαιροποίησης και να είναι ε, διαθέσιμα για τους διδάσκοντες. Νομίζω ότι αυτό είναι το στίχημα που έχουμε να απαντήσουμε. Αυτό επίσης που είναι σημαντικό είναι, και αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε, είναι να επαληθεύσω με των καλύτερων εμπειριών που υπάρχουν, τις βέλτιστες πρακτικές που έχουμε στα κράτη-μέλη, οι οποίες ε, ε, αναφέρονται και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι βέλτιτες πρακτικές ε, και από αυτά τα κέντρα που μας έλεγε προηγουμένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που γεννήθηκαν από το πρόγραμμα Safer Internet που θεωρώ ότι είναι μία από τις σημαντικότερες πτυχές είναι λοιπόν ένα πραγματικό δίκτυο πλέον που ε, προχωρά και αποτελεί κίνητρο και για τα κράτη-μέλη αλλά και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δημιουργήσουν όχι μόνο νέα νομοθεσία αλλά και νέες συμφωνίες. Ακόμα και η συμφωνία που προωθεί η Νέλη Κρούς ε, προκύπτει από αυτό το κίνητρο που έχει δημιουργηθεί από αυτό το ευρωπαϊκό σύστημα και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον διότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι καλύτερες ε, λύσεις προκύπτουν μέσα από συμμαχίες. Η ισχύς εν το και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό θα βρούμε έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα τα οποία δεν είναι δημόσια αγαθά. Για παράδειγμα, η παραβίαση, η παραβίαση της ταυτότητας και της εικόνας των παιδιών που χρησιμοποιούνται από εκεί και πέρα για τα προφίλ όπως αποκαλούνται από την κοινωνία και ούτε καθεξής για να χρησιμοποιηθούν Ε, τα στοιχεία τους. Ε, επομένως, παιδιά που ανεβάζουν στοιχεία στο διαδίκτυο ε, δεν θα μπορούν πια να τα σβήσουν. Ακόμα και συζητήσεις για το σεξ, φωτογραφίες τους δεν θα μπορούν να διαγραφούν ακόμα και όταν είναι ενήλικες. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε μια ισορροπία και να συμπεριλάβουμε στην έκθεση και ότι έχουμε από πλευράς νομοθεσίας αλλά και από πλευράς εκπαιδευτικών συμμαχιών, συμμαχιών αν θέλετε ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να τονίσουμε όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία των ανηλίκων όλα αυτά υπό ένα πρίσμα που θα λαμβάνει υπόψη όπως έλεγε προηγουμένως και ο κύριος Φοντάνα, το γεγονός ότι υπάρχει τόσο γρήγορη εξέλιξη και είναι τόσο διαφορετική η προσέγγιση παιδιών ε, σε νέες μορφές επικοινωνίας που δεν μπορούμε να τα ε, ε, απαγορεύσουμε ε, στο όνομα μιας υπερβολικής ανησυχίας, αλλά ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και τα θέματα της παιδικής πορνογραφίας, ακόμα και στις πιο ήπιες μορφές του, που εκμεταλλεύεται την ψυχολογία των παιδιών. Ελπίζω λοιπόν με τη βοήθειά σας να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια καλή έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Hey, thank you, Mrs. Costa. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Υπανορισμένοι για το θέμα αυτό ότι είναι πολύ πιο εύκολο να συζητήσουμε για τους στόχους και όχι για τα μέσα. Θα υπάρξουν πολλές συζητήσεις για τα θέματα αυτά και είναι τμήμα του γενικού θέματος της εφιούς και κατάλληλης ρύθμισης στο διαδίκτυο και όπως βλέπετε και με τη συζήτηση για τη Συμφωνία Άκτα δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Έχουμε λοιπόν την παρουσίαση του σχεδίου έκθεση της 25 Απριλίου και θα ψηφίσουμε και θα εγκρίνουμε την έκθεση της κυρίας Κώστα στις 20 Ιουνίου. Πάμε στο επόμενο θέμα, το θέμα 13, κοινέ ρυθμίσεις για, τους Ευρωπα... για τα Ευρωπαϊκά Διεθνωτικά Ταμεία και κατάργηση κανονισμών. Η κυρία Μπεναράπ Ατού είναι η συγγήτρια για τα δύο αυτά θέματα, δύο νομοθετικές ε, γνωμοδοτήσεις για την ε, Περιφερειακή Επιτροπή και για την Επιτροπή Απασχόληση. Καταρχήν, κοινέ διατάξει για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ο στόχο είναι να έχουμε ένα κοινό πλαίσιο κανόνων για την επόμενη περίοδο 2014-2020 των διαφθορτικών πόρων. Θεσπίζει βασικές αρχές για γενικές ε, αρχές υποστήριξης όπω είναι εταιρική σχέση, πολυμερής ε, διακυβέρνηση, ισότητα ανδρών και γυναικών, αυτή είναι λοιπόν οι βασικές αρχές των νέων προτάσεων για τους διαφορετικούς πόρους που θα καλύψουν το 1 τρίτο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι βασικά στοιχεία επίδοξης της στρατηγικής της Ευρώπης 2020. Η Επιτροπή Περιφερειών θεμάτων είναι, Περιφερικών Θεμάτων είναι η επί της ε, αρμόδια και δίνω τώρα το λόγο στη Μαλίκα. Ευχαριστώ, Άλιο. Όπως το υπενθύμισες, η Κομισιόν στο 6 Οκτωβρίου του 2011 υιοθέτησε ένα σύνολο νομοθετικών προτάσεων για την πολιτική συνοχή της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2014-2020. Ε, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να τις εξετάσουν προκειμένου να υιοθετηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου του 2012. Η εργασία αυτή είναι σημαντική διότι στα διευθυντικά ταμεία αφιερώνεται περίπου το 1 τρίτο του συνολικού προπολογισμού για την περίοδο 2007-2013, το 35% συνολικά συγκεκριμένα. Και είναι μετά τη Γεωργία το δεύτερο μεγαλύτερο έξοδο, η δεύτερη μεγαλύτερη δαπάνη του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, τα χρηματοδοτούνται ε, πολύ άριθμα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αυτών των μοσών. Η διαφορετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι η μεγαλύτερη ε, συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικά μας θέματα του πολιτισμού. Για να βγούμε από την Ευρώπη της κρίσης, τα μέτρα λιτότητας δεν αρκούν το υπενθυμίσαμε και χτες και προχτές, συζητώντας το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Μόνη τη η δεν δίνει τη λύση. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν όλα τα εργαλεία που διαθέτουμε μέσω αυτών των ταμείων για μια πιο ισόρροπη προσέγγιση, για να προωθήσουμε την οικονομική συνοχή, ε, αλλά ταυτόχρονα και την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Ο ρόλος των διαχρονικών ταμείων ε, είναι αυτός ακριβώς, πρέπει να είναι ευέλικτα, να έχουν τους κατάλληλους πόρους και να ανταποκρίνονται στις ε, ανάγκες των πολιτών. Σε ό,τι αφορά τις κοινέ διατάξεις, η Κομισιόν ε, προτείνει στο εγγραφό της κάποιες τροποποιήσεις. Οι δύο πιο σημαντικές αφορούν και είναι θετικέ αλλαγές πιστεύω. Η πρώτη αφορά την απλοποίηση των εφαρμοστέων κανόνων. Θα υπάρχει πλέον ένα σύνολο κανόνων για όλα τα ταμεία και θα ακολουθείτε μια πιο ενιαία προσέγγιση για να ε, απομακρυνθούμε από τη σημερινή κατάσταση που έχουμε διαφορετικούς κανόνες για κάθε ταμείο. Οι στόχοι των ε, ταμείων ε, μέσω αυτών των κανόνων θα είναι επίσης πιο συνεκτικοί και προφανώς πιο αποτελεσματικά θα επιτυγχάνονται. Δεύτερη μεγάλη αλλαγή προτείνει η Κομισιόν είναι η συγκέντρωση της χρηματοδότησης σε ένα περιορισμένο αριθμό στόχων. Θεματική λοιπόν εστίαση, ε, στόχοι οι οποίοι θα συνδέονται προφανώς με τη στρατηγική 2020 που έχει ως στόχο την ευφυή, βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. Αυτές οι αλλαγές, αυτή η αλλαγή είναι πολύ θετική γιατί αφορά ιδιαίτερα την εκπαίδευση, την παιδεία, μας αφορά λοιπόν την κατάρτιση, την κοινωνική συμπερίληψη και προφανώς αφορά άμεσα τις αρμοδιότητές μας. Παρόλο ότι το κείμενο ε, αναφέρεται σε γενικές ε, ε, διατάξεις και τεχνικές διατάξεις, το περιεχόμενο μας αφορά ιδιαίτερα και θα πρέπει να εξετάσουμε ιδιαίτερα ορισμένα πράγματα όπως τον τίτλο 2, τον σχετικό με τη στρατηγική προσέγγιση, καθώς επίσης και το παράρτημα 4 σχετικά με τις ε, με την αιρεσιμότητα και, τις, ε, ε, τις, τους εξάν, εξάντε προϋποθέσεις. Τώρα, για το κοινωνικό ταμείο, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η πρόταση κανονισμού είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί μεταξύ των βασικών θεμάτων ε, είναι η πρόθεση της απασχόλησης, ε, η επαγγελματική κινητικότητα, η επένδυση στην εκπαίδευση, ε, την κατάρτιση διαβίου, διαβίου κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την καταπολέμηση της φτώχειας. Ε, συνδέεται με τη στρατηγική για την ε, απασχόληση και τις ε, νέες δεξιότητες, την πλατφόρμα εναντίον της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη στρατηγική για την ψηφιακή Ευρώπη και τις πρωτοβουλίες για την Ευρώπη της καινοτομίας. Δεύτερον, γίνονται, γίνεται ιδιαίτερη πρόοδος στα εξής θέματα. Άρθρο 3, πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, βλέπουμε ότι συμπεριλαμβάνεται και η μείωση της πρόορης εγκα... σχολικής εγκατάλειψης που μας αφορά ιδιαίτερα και, την... και η πρόθεση της ε, πρόσβασης σε σε προσχολική ε, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η απασχόληση των ε, νέων και η υποστήριξη ε, των περιθωριακών ομάδων και των λιγότερο προνομίχων ομάδων είναι επίσης συστήματα του στόχου. Το 20% του προπολογισμού θα αφιερωθεί στην καταπολέμηση της φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού και τρίτον, ε, άρθρο 9, ε, ιδιαίτερα τονίζεται η κοινωνική καινοτομία. Θα πρέπει βέβαια να οριστεί καλύτερα αυτό ο όρο. Τι ακριβώ σημαίνει κοινωνική καινοτομία, Σω θα πρέπει να το ορίσουμε καλύτερα στο κείμενο. Ε, Εμεί εργαζόμαστε πολύ καιρό σε αυτά τα θέματα Ε, μην ξεχνάμε τη γνωμοδότηση τη κυρία ε, Κώστα για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αντίον τη Φτώχεια και την έκθεση τη κυρία Σόνεμπουλ για την ε, μείωση τη ε, πρόορη κατάληψη τη σχολική εκπαίδευση. Όμω μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη γνώμη μα, τι νομοδοτήσει μα και να εστιάσουμε στι δικέ μα προτεραιότητε. Έχω όμω και κάποιε επιφυλάξει σε ό,τι αφορά αυτέ τι αλλαγέ προτείνει η Κομισιόν. Καταρχήν, ορισμένε διατάξει του κανονισμού 2007-2013, του ισχύοντος κανονισμού δηλαδή, ε, περιελάμβαναν κάποια στοιχεία τα οποία πλέον δεν εμφανίζονται στι καινούργιε προτάσει κομισιών. Το ε, έκτο εδάφιο τη ε, έκθεση, που αναφέρεται στο πρόγραμμα Equal για παράδειγμα ε, πολέμηση ε, των ανισοτήτων στο χώρο εργασίας που δεν εμφανίζεται πλέον στην καινούργια έκθεση, καινούργια πρόταση. Επίση, το άρθρο 3 του ισχύοντο κανονισμού για την κοινωνική συμπερίληψη που αναφέρεται ιδιαίτερα στην ε, επαγγελματική κατάρτιση και στην εκπαίδευση που επίσης δεν βλέπουμε στο καινούριο κείμενο. Ο πολιτισμό επίση δεν αποτελεί στόχο προτεραιότητα, παρόλο που συνδέεται άμεσα με την εκπαίδευση, την κοινωνική συμπερίληψη και την καινοτομία. Δηλαδή, που είναι στόχοι τη στρατηγική 2020. Συνεπώ, θα πρέπει να είμαστε λογικά συνεπεί. Θεωρώ ότι η πολυεπίπεδη ε, συνεισφορά του πολιτισμού στην οικονομική ανάπτυξη, στην κοινωνική συμπερίληψη, ε, στην κοινωνική ένταξη των περιφερειακών ομάδων δεν, ε, ομάδων δεν αναγνωρίζεται επαρκώς. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ρητά ότι τα σχέδια τα project που έχουν ε, πολιτιστική διάσταση θα πρέπει να συμπεριληφθούν και γι' αυτό λόγο θα πρέπει να γίνει μια προσθήκη στο άρθρο 3. Τελειώντας να πω τα εξής. Πρόκειται για σημαντικά ποσά, σημαντικά κονδύλια. Ελπίζω ότι η συζήτηση θα ε, είναι καρποφόρα και σας ευχαριστώ ήδη εκ των προτέρων για τη ε, συνεισφορά σας. Ευχαριστώ Μαλίκα. Ο κύριος Μπόρις ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μπόρης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπούμε σε περισσότερο βάθος στο κείμενο του κανονισμού, να το αναλύσουμε λεπτομεριακά. Να δούμε καταρχήν ποια είναι η τωρινή δημοσιονομική πρόβλεψη. Προφανώς εκπνέουν οι τωρινές δημοσιονομικές προοπτικές, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις μελλοντικέ προτάσεις, γιατί η στρατηγική της Ευρώπης 2020 είναι κεφαλαιόδου σημασία. Το θέμα της απλοποίησης είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλούς και ιδίως τους αποδέκτες αυτών των ταμείων και πάντα για τον πολιτιστικό τομέα ένα βασικό πρόβλημα είναι ο αποκλισμός από την μελλοντική περίοδο προγραμματισμού επενδύσεων σε τομείς πέραν θεμάτων ε, πολιτιστικής κληρονομιάς κτλ. Αν κάποιος θέλει να, δημιουργήσει ένα σύγχρονο μουσείο, αν θέλει να ψηφιοποιήσει κινηματογραφικές ταινίες, Κάτι λοιπόν που δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, που δεν έχει ηλικία 100 ετών. Σύμφωνα με τις νέες πρότασεις δεν μπορούν να δοθούν χρηματοδοτήσεις για τέτοιες επενδύσεις. Αντί να δίνουμε λοιπόν επενδύσεις για την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών στο υψηλότερο επίπεδο, εμείς κάνουμε κάτι που είναι ουσιαστικά το αντίθετο. Μιλάμε για εκπαιδευτική δραστηριότητα στον πολιτιστικό τομέα, αλλά από αυτά τα οποία ακούσαμε και είδαμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας δίνει καμία απολύτως εγγύηση σε σχέση με το πρόγραμμα «Η νεότης σε δράση». Δεν μας εγγυάται ότι κάποια προγράμματα θα εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούνται στο μέλλον. Ο έρασμος για όλους και άλλα προγράμματα, ακόμα και αυτά είναι υπό απειλή. Οι νέες αυτές προτάσεις λοιπόν είναι μια απειλή για τον πολιτιστικό τομέα και για προγράμματα στο τομέα αυτό που έχουν αποδειχθεί επιτυχίες. Κυρία Σάντς, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να επανέλθω σε ορισμένα σημεία που ανέφερε η Μαλίκα, που μπήκε στην ουσία του θέματος. Υπάρχουν πολλές νέες προτάσεις στο πακέτο αυτό. Ο στόχος είναι μεγαλύτερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη αποδοτικότητα, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και ερεσιμότητα για μια πολιτική συνοχή για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα επάγρυπνοι για ορισμένα θέματα, ιδίως για, για τη συγκέντρωση σε ορισμένους θεματικούς τομείς προτείνει 11 προτεραιότητες αυτός ο κανονισμός από τις οποίες θα πρέπει να επιλέξουν οι περιφέρειες της Ευρώπης. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτό το οποίο λαμβάνει η Κομισιόν, η παιδεία και η εκπαίδευση δεν έχουν σημαντικό ρόλο και δεν εμφανίζονται με προφανή τρόπο μέσα σε αυτήν την κατανομή σε θεματικούς τομείς. Επιπλέον η Κομισιόν στις προτάσεις της θέλει να επιβάλλει ε, να δοθεί το μεγαλύτερο ημερίδα του λέοντος αυτών των πόρων στην προστασία του περιβάλλοντος. Βλέπουμε σήμερα στα κονδύλια του Περιφερειακού Ταμείου τα πολιτιστικά θέματα να είναι μία από τις προτεραιότητες των περιφερειών της Ευρώπης στα λειτουργικά τους προγράμματα. Θα πρέπει εμείς να ζητήσουμε να εφαρμοστεί υποχρεωτικά ένα ποσοστό για τις επενδύσεις στον τομέα της κουλτούρας και της παιδείας. Είναι απαραίτητο να προωθήσουμε την κατάρτιση και την ε, κοινωνική συμπερίληψη με την υποστήριξη της ε, παιδείας και του πολιτισμού. Ευχαριστώ πολύ, λέει Ο κύριος Μάτουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη δική μου πλευρά θέλω να κάνω ορισμένε παρατηρήσεις για τον κανονισμό αυτόν ο οποίος προτείνεται. Όπως ελέγχθη ήδη προηγουμένως, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα θέματα αυτά, ότι δηλαδή ο νέος αυτός κανονισμός έχει σαν εκπεφρασμένο στόχο μία απλοποίηση όλων των κανόνων, αλλά συγχρόνως οδηγεί και σε μια συγκέντρωση των στόχων. Αυτή η συγκέντρωση των στόχων έχει όμως κάποιες επιπτώσεις. Στην πράξη σημαίνει ότι διαγράφεται η τάση, οι πόροι αυτοί να χρησιμοποιούνται, να χρηματοδοτούν μόνο προγράμματα μεγάλης εμβέλειας. Εμείς στην Επιτροπή μας Ξέρουμε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα προγράμματα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, του πολιτισμού, της παιδείας. Ξέρουμε ότι ακόμα και με μικρά ποσά μπορούμε να κάνουμε ορατά τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών. Αυτή τη στιγμή ο κίνδυνος είναι όλα αυτά τα μικρά μέσα σε εισαγωγικά προγράμματα δεν θα χρηματοδοτούνται στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ επάγρυπνοι στην Επιτροπή μας να βρούμε λύσεις ώστε τα προγράμματα αυτά στον τομέα του πολιτισμού να συνεχίσουν να υπάρχουν και να είναι επιλέξιμα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη θεματική συγκέντρωση και τον περιορισμένο αριθμό των στόχων, εγώ θέλω να υπενθυμίσω και μια άλλη πτυχή του προβλήματος αυτού. Οι ευρωπαϊκές περιφέρειες είναι πολύ Είναι πολύ δύσκολο να μπορούμε να βάλουμε στο ίδιο καλούπι δύο περιφέρειες διαφορετικές ακόμα και σε μία και την αυτή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κίνδυνος λοιπόν της υπερσυγκέντρωσης στο θεματικό τομέα οδηγεί σε προβλήματα. Θα ήταν καλύτερο η απόφαση να λαμβάνεται σε πιο αποκεντρωμένο επίπεδο, όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη. Ελπίζω στην Επιτροπή Πολιτισμού θα βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση, ώστε να κρατήσουμε αυτά τα προγράμματα που μας ενδιαφέρουν. και ευχαριστώ την εισηγητή για όλα αυτά που μας παρουσίασε σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Μάτουλα. Κάποιος άλλος θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ή τότε θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να λάβει το λόγο. Είσαστε έτοιμοι. Παρακαλώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ. Ρέιτσι Λάγκρι από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή Πολιτική, Θα ξεκινήσω λοιπόν απαντώντα κάποια θέματα για τον κανονισμό για τι κοινέ διατάξει, και από εκεί και πέρα ο συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση, θα απαντήσει στα θέματα που αναφέρονται στον κανονισμό για το Κοινωνικό Ταμείο. Γιατί λοιπόν θα μιλήσουν δύο από εμά ε, μια σύντομη εξήγηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά τα θετικά λόγια της εισηγήτριας. Προσπαθήσαμε να απλουστεύσουμε ε, τα θέματα αυτά και η απλούστευση να αποτελέσει ορόσημο της όλης μας ε, πολιτικής. Ε, όσον αφορά τη θεματική συγκέντρωση άκουσα κάποια θετικά στοιχεία αλλά και κάποια ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο προωθείτε. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να ακούμε και τα καλά σας λόγια ε, στο μέλλον θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό της χρηματοδότησής μας. Όπως γνωρίζετε, πολλές από τις ε, επικρίσεις της ε, πολιτικής συνοχής στο παρελθόν είχαν σχέση με το γεγονό ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να πλώσουμε τόσο λεπτή φέτα, κομμάτι βούτυρο στη φέτα του ψωμιού που δεν υπάρχει καμία γεύση πλέον. Αυτό είναι σαφές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στην ευρύτερη επικράτεια. Γι' αυτό λοιπόν στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να έχουμε πολιτικές που θα έχουν τις μέγιστες δυνατές ε, επιπτώσεις αλλά και συμβολή. Τι προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε με αυτούς τους θεματικούς στόχους. Όπως αναφέρθηκαν από την εισηγήτρια, προέκυψαν σαφώς από το Ευρώπη 2020 που είναι η στρατηγική που συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από όλους τους φορείς προκειμένου να μας βοηθήσει να ε, ε, ε, διαφύγουμε τις κρίσεις και να έχουμε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο προέκυψαν οι θεματικοί στόχοι. Και από εκεί και πέρα, βάσει του κανονισμού, είδαμε συγκεκριμένε επενδυτικέ προτεραιότητες βάσει κάθε ταμείου. Αλλά ε, δεν παρεμβαίνουν στην επιλεξιμότητα των παρεμβάσεων. Και γι' αυτό θα ήθελα τώρα εδώ να σας πω κάποια πράγματα για τον κανονισμό η e ERDF ε, για το Περιφερειακό Ταμείο λοιπόν, ε, διότι αναφέρθηκαν ε, τα θέματα της επιλεξιμότητας από κάποιους ομιλητές και προτείνουμε να επικεντρωθούμε στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, διότι θεωρούμε ότι αυτά θα πρέπει να κάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για να επιτύχουμε τους στόχους του Ευρώπη 2020. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε σε κάθε περιφερειακή περιφέρεια πόσο θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάθε θεματική ενότητα, αλλά σε αυτά θα πρέπει να σταθούμε. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν αποκλείεται. Μπορεί να εμπίπτει σε κάποιον από αυτού του στόχου. Για παράδειγμα, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι πολύ σημαντικό ε, παράγον τη ε, πολιτιστική κληρονομιά. Οπότε μπορεί να δείτε κάτι για την πολιτιστική κληρονομιά που να συμμετέχει στην ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, το ίδιο μπορούμε να έχουμε σε άλλο θεματική ενότητα Ω ως επενδυτική προτεραιότητα για την πολιτιστική κληρονομιά. Δηλαδή, οι θεματικέ ενότητε δεν είναι ισοδύναμε τη επιλεξιμότητα. Τα προγράμματα ε, δεν είναι μη επιλέξιμα γιατί δεν αναφέρονται συγκεκριμένα ω θεματικέ ενότητε. Να πω τώρα ότι εκ των προτέρων ερεσιμότητα είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας είπατε. Περιμένουμε να δούμε τι θα μας πείτε κυρία Συγήτρια στην έκθεσή σας. Ε, τώρα, για όλους τους παρισταμένους να πω ότι ο λόγος που το έχουμε συμπεριλάβει το στοιχείο αυτό είναι για να είμαστε βέβαιοι στο μέτρο του δυνατό ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι όροι για να επιτύχουμε. Αυτό που είδαμε πολλές φορές με τη χρηματοδότηση στις πολιτικές στο παρελθόν είναι ότι είτε το πλαίσιο της πολιτικής, είτε το ρυθμιστικό πλαίσιο, είτε το θεσμικό πλαίσιο δεν ε, ήταν επαρκή. Για παράδειγμα, είχαμε χρηματοδότηση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά χωρίς στρατηγική για το πώς μπορούμε να έχουμε εφαρμογή στη συγκεκριμένη περιφέρεια περιφέρεια ή σε άλλες δυνατότητε χρηματοδότησης. Προσπαθούμε λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τους κατάλληλου όρου για να επιτύχουμε. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης για να μιλήσει για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος και δίνει το λόγο στον συνάδελφο της κυρίας. Καλημέρα. Διαβάζω στη, ε, δουλεύω στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Ε, θα σχολιάσω αυτά τα οποία ελέγχθηκαν και τις ε, παρατηρήσεις, τις επιφυλάξει που εκφράστηκαν για το θέμα του Ευρωκοινωνικού Ταμείου και σε σχέση με την, τον πολιτισμό. Ο, η αποστολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου, όπως ορίζεται από τη συνθήκη, είναι η βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης, της απασχολησιμότητας δηλαδή των Ευρωπαίων εργαζομένων. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή που καθορίζεται από τη συνθήκη επαναλαμβάνω και την οποία υπενθυμίζουμε και εμείς στην πρόταση κανονισμού μας. Αυτή η αποστολή ε, είναι και η βάση όλων αυτών των προτάσεων που κάνουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνεισφέρει σε τρεις ε, από τους βασικούς στόχους της ε, στρατηγικής ε, Ευρώπη 2020 απασχόληση, παιδεία και κοινωνική συμπερίληψη και καταπολέμηση της φτώχειας. Το πεδίο εφαρμογή που προτείνεται στο άρθρο 3 ακριβώς επαναλαμβάνει αυτούς τους τρεις στόχους. έχει ένα πρώτο θεματικό στόχο την απασχόληση, ένα δεύτερο την ε, παιδεία και έναν τρίτο την κοινωνική συμπερίληψη και την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε σχέση με τον τρέχοντα κανονισμό ενισχύουμε πλέον την προτεραιότητα της ε, παιδείας και του τρίτου άξονα, δηλαδή της καταπλήνωσης της φτώχειας και της κοινωνικής υπερήλυψης... Έχοντας στο μυαλό μας βέβαια τους στόχους της Ευρώπης 2020. Ο πολιτισμός αυτός καθ' αυτός δεν αναφέρεται στου στους θεματικούς άξονες αλλά συνδέεται άμεσα και στενά με τον θεματικό άξονα της παιδείας. Όπως το υπενθύμησε και η Ρέιτσελ, οι θεματικοί άξονες δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα θέματα επιλεξιμότητας και με τα project, τα, οποία, τα σχέδια τα οποία θα υλοποιηθούν ε, και θα έχουν σχέση με την παιδεία. Project που θα, έχουν, που θα εντάσσονται σε έναν από αυτούς τους τρεις ε, θεματικούς άξονες ε, θα μπορούν να εγκριθούν και προφανώς θα μπορούν να αγγίζουν και τα σχετικά με, την, με τον πολιτισμό. Τώρα, απουσία αναφοράς του προγράμματος Equal στην αιτιολογική έκθεση, τα εκτιμώντας. Το Equal ήταν ένα ε, κοινοτικό εργαλείο της περίοδου 2020. Το είχαμε συμπεριλάβει στην αιτιολογική έκθεση του τρέχοντος, ισχύοντος κανονισμού προκειμένου να οθήσουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους ε, τα διδάγματα που προέκυψαν από την υλοποίηση του Equal στα επιχειρησιακά τους προγράμματα. Αυτό το ονομάζουμε mainstreaming συνήθως. Αυτό το mainstreaming ε, είχε ε, μια ε, επιτυχία σχετική, διαφορετική σε κάθε κράτος μέλος. Οι αρχές, οι βασικές αρχές της πρωτοβουλίας Equal είναι ήδη πολύ παρούσες την πρόταση που κάνουμε για τον κανονισμό του Κοινωνικού Ταμείου. Για παράδειγμα, η ε, σύμβαση σύμπραξη, η ισότητα, η αρχή της μη διάκρισης, της αποφυγής των διακρίσεων, ε, πράγματα στα οποία το equal συνεισέφερε πάρα πολύ. Θα τελειώσω αναφέροντάς σας την σύνδεση με άλλα κοινωτικά εργαλεία, το Erasmus, η πρωτοβουλία νεότητα σε κίνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, μεταξύ των θεματικών του στόχων, έχει και την κινητικότητα, την πρόθεση της κινητικότητας. Απασχόληση και κινητικότητα. Συνεπώς, η πρόταση της Κομισιόν συμπληρώνει τα υπάρχοντα εργαλεία, έρασμους και νεότητα σε κίνηση. Δεν θέλουμε να τα αντικαταστήσουμε, αλλά να τα συμπληρώσουμε. Ήδη ακόμα και σήμερα, ορισμένα κράτη χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για δράσεις κινητικότητας παρόμοιες με αυτές που χρηματοδοτεί το έρασμος. Όταν θεωρούν τα κράτη-μέλη ότι χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση, χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Ε, Μαρίκα, Ευχαριστώ, Μαρίκα. Θες να πεις κάτι? Θέλω απλώ να σα υπενθυμίσω το πρόβλημα το οποίο τίθεται για το γεγονό ότι σε κάποιε περιφέρειες δεν υπάρχει η επαρκή απορρόφηση του, των πόρων του κοινωνικού ταμείου, ακόμα και σε μια χώρα όπως η Ισπανία που βρίσκεται σε κρίση και που το κοινωνικό ταμείο είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίσει την κρίση, η Ισπανία δεν χρησιμοποιεί όλα τα κονδύλια του κοινωνικού ταμείου. Τι λύση θα μπορούσατε να θέσετε για το θέμα αυτό, να προτείνετε για το θέμα αυτό. Είναι μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Παρακαλώ. Είχαμε προβλήματα απορρόφησης τα πρώτα χρόνια που δεν ήταν ε, αμεληταία. Πάρα πολλά ταμεία έχουν προβλήματα στο επίπεδο απορρόφησης των πόρων, αλλά σιγά σιγά βελτιώνεται η κατάσταση αυτή. Είναι υψηλότερο το επίπεδο απορρόφησης, γιατί στο τέλος του 2000... 2012 λέει ο μιλητής, 2011 εννοεί, ε, είχαν ε, ε, εξαντληθεί όλοι οι πόροι για πιστώσεις πληρωμών και χρειάστηκε να μεταφέρουμε, να καθυστερήσουμε ορισμένες πληρωμές. Για την περίπτωση της Ισπανίας, χωρίς να πω σε λεπτομέρειες, <clears throat> υπήρξαν κάποια προβλήματα για την εφαρμογή συστημάτων που τροχοπέδησαν σημαντικά την εφαρμογή του, την ε, εφαρμογή προγραμμάτων και τις πληρωμές επί το οποίο δεν μπορώ να σας δώσω λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά αλλά η Γενική Διεύθυνσή μας έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό που ήταν τεχνικού χαρακτήρα και που εμπόδισαν μια μεγάλη απορρόφηση των πόρων του Κοινωνικού Ταμείου στην Ισπανία. Αλλά μπορώ να επανέλθω σε εσά για να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες αν επιθυμείτε. Κύριε Μαρές, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς να προσθέσω μια πληροφορία που νομίζω ότι είναι σημαντική ότι αποφάσισε στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αποστελούν αποστολές σε 8 χώρες όπου υπάρχει μεγάλη ανεργία. Μια αποστολή στην Ισπανία που είναι πριν από δύο μέρες και τις οποία ο κύριος στόχος ήταν να δει πώς πηγαίνει η χρήση των διαδοτικών πόρων και ιδιαίτερα του Κοινωνικού Ταμείου για να ανακατευθύνουμε τους πόρους αυτούς σε δράσεις υπέρ της καταπολέμησης ανεργίας των νέων και ή δυνατόν να τους ε, παρακινήσουμε να μπουν στα προγράμματα Εράσμος ή Λεωνάδο. Ωραία. Τότε, τον Απρίλιο, έχουμε την εξέταση του σχεδίου έκθεσης και θα επανέλθουμε. Προχωρούμε στο σημείο 15 στη μέση διάταξη. Είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση και Ευρώπη 2020. Η κυρία Χάνιμπολ είναι συγήτρια. Ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Χάνιμπολ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση για την οποία θα κάνουμε τώρα την πρώτη ανταλλαγή απόψεων είναι απάντηση σε κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου για την εφαρμογή του στρατηγικού έργου για την ε, ευρωπαϊκή συνεργασία για την εκπαίδευση και την κατάρτιση που είναι και αυτό στην στρατηγική Ευρώπη 2020. Έχουμε πάρα πολλά 2020 και θα προσπαθήσω να καταστήσω σαφές για ποιο 2020 μιλάω εγώ. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολογεί πού βρισκόμεθα όσον αφορά την εφαρμογή της ε, ε και κατάρτισης το 2020 δεδομένων και των οικονομικών συγκυριών ε, που επηρεάζουν πολύ και τις αποφάσεις που λαμβάνουμε αυτή τη στιγμή. Πολύ πριν γίνει τόσο δύσκολη οικονομική κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή, το Συμβούλιο ετοίμασε το στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ε, που είναι το πρόγραμμα του 2020, αλλά έκτοτε το πλαίσιο έχει αλλάξει και αντιμετωπίζουμε νέες αβεβαιότητες και περιορισμούς ως Ευρωπαϊκή Ένωση και ως κράτη-μέλη σε κάποιες περιπτώσεις υποχρεωθήκαμε να λάβουμε κάποια μέτρα ώστε να αντιμετωπίσουμε την χείριση χειρότερη οικονομική κρίση που αντιμετωπίσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, στην ιστορία της Ευρώπης ε, τον τελευταίο αλλά και τον προηγούμενο αιώνα. Συμφωνήσαμε λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι χρειαζόμαστε μία στρατηγική για ευφυή, βιώσιμη ε, ανάπτυξη η οποία είναι γνωστή ως Ευρώπη 2020. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, κάτι το οποίο είναι θετικό, διότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση πλέον αναγνωρίζονται ως ζωτική σημασία για την οικονομία μας, για τη λειτουργία της οικονομίας και για τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας για το μέλλον. Υπάρχουν ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές και εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης και συγκεκριμένες συστάσεις αναχώρα που είναι γνωστές ως CSR και θα έπρεπε να αποτελούν οδηγό για τις μεταρρυθμίσεις των κρατών μελών. Έναν από τους πέντε στόχους για το 2020 αφορά ε, την πρόορια κατάληψη του σχολείου ε, σας έχω αναφέρει το ζήτημα αυτό και στο παρελθόν. Υπήρχε και σχετική έκθεση, αλλά όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ε, δεξιότητες και τα επιτεύγματα, ε, το να ολοκληρώνει κάποιος τη σχολική του εκπαίδευση σημαίνει ότι μπορεί μακροπρόθεσμα να έχει καλύτερες θέσεις εργασίας. Είναι λοιπόν ένας στόχος τον οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουμε σε οποιαδήποτε αξιολόγηση της, της οικονομικής κατάστασης και οποιαδήποτε στρατηγική για να λάβουμε μέτρα. Βέβαια δεν είναι όλα τα θετικά τα στοιχεία και υπάρχει ένα ποσοστό μικρότερο του 15% το να έχουμε ε, ένα στόχο λοιπόν ε, που να εγκαταλείπουν το σχολείο σε ποσοστό μικρότερο του 15% καταλαβαίνετε ότι ο στόχος αυτός είναι πολύ δύσκολος έχουμε λοιπόν αυτούς τους στόχους που προσπαθούμε να επιτύχουμε ε, και πρέπει να τους έχουμε κατά νου η οικονομική κρίση επηρεάζει σαφώς τις προοπτικές των νέων ανθρώπων. Η ανεργία των νέων κυμαίνεται από το 15,5% το 2008 που ήταν ήδη πολύ ψηλή στο 20,9% το 2010 που είναι τεράστιος αριθμός. Πρόκειται για ένα πέμπτο νέων ανθρώπων χωρίς θέση εργασίας και ε, υπάρχει ένα μερίδιο 18 ε, έως 24 ετών που δεν είναι ούτε σε διαδικασία εκπαίδευσης, ε, ούτε έχουν θέση εργασίας αυτή τη στιγμή, ούτε λαμβάνουν κάποια κατάρτιση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να παραμένουν οι νέοι άνθρωποι στο σχολείο και να γνωρίζουν τι συνέπειε έχουν να αντιμετωπίσουν αν εγκαταλείψουν το σχολείο πολύ νωρί. Ο στόχο του Ευρώπη 2020 είναι να μειωθεί αυτό το μυρίδι τη ομάδα των 18-24 ετών που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο στο ένα ποσοστό κάτω του 10% μέχρι το 2020. Ε, Βεβαίω αυτό ο στόχο στα πλαίσια και τη οικονομική κρίση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει ωστόσο να γνωρίζουμε ότι αν συνεχίσουν οι τάσει τάσεις ε, και τα στατιστικά στοιχεία που σα έδωσα συνεχίσουν σε αυτά τα επίπεδα ή επιδεινωθούν, δεν θα επιτύχουμε του στόχου αυτού. Επομένω, προκειμένου να ε, αναδειχθούμε ισχυρότεροι από αυτή την κρίση, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ανάπτυξη. Και εδώ νομίζω έρχεται και ο ρόλο τη επιτροπή μα και αυτό που κάνουμε στην Επιτροπή μας ε, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Διότι ένα από του τρόπου με του οποίου θα δημιουργήσουμε ανάπτυξη είναι μέσω τη γνώση και τη καινοτομία. Και η ανώτατη εκπαίδευση είναι προφανώς ο δρόμος και ο κινητήριος μοχλός προς αυτό το σκοπό. Η ανώτατη εκπαίδευση μπορεί να παράσχει ένα εργατικό δυναμικό υψηλών δεξιοτήτων, δυναμικό το οποίο χρειαζόμαστε για να έχουμε ανάπτυξη και εξέλιξη και για να δώσουμε τα εφόδια που χρειάζονται όλοι σε αυτή την ε, εντατική αγορά εργασίας. Πρέπει να εξετάσουμε και τα θέματα της διαβίου μάθησης και θα πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές επ' αυτού η διαβίου μάθηση υπό την έννοια του, της συνεχούς εξέλιξης στη διάρκεια της ζωής σου δεν ισχύει στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα πρόσφατα στοιχεία για αρκετούς ενήλικες ε, ηλικίας 25 έως 64 για τη συμμετοχή του στη διαβίου μάθηση καταδεικνύουν ότι μειώνεται η διαβίου μάθηση παρά τις προσπάθειες και τις καλές πρωτοβουλίες που είχαμε. Δυστυχώς το χάνουμε το παιχνίδι. Ε, αυτή τη στιγμή Έχουμε ένα στοιχείο για το 2010, δεν έχω στοιχεία για αργότερα, 9,1% ε, ε, του ενεργού πληθυσμού συνεχίζουν στη διαβίου μάθηση και είναι πολύ πιο χαμηλό από το στόχο του ε, Ευρώπη 2020, διότι δηλαδή θέλουμε να έχουμε ένα 15% μέχρι το 2020. Υπάρχουν λοιπόν άνεργοι νέοι και ενήλικες οι οποίοι δεν εξελίσσουν περαιτέρω τις δεξιότητές τους. Αυτό λοιπόν μας ε, οδηγεί προς το συμπέρασμα ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν οι επενδύσεις που θα έπρεπε να υπάρχουν, επενδύσεις σε δεξιότητες και εδώ εμείς αν θέλουμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν ανάπτυξη και να έχουμε συνεχή εκπαίδευση αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε θέσεις εργασία μέσω οικονομικής ανάπτυξης και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε τη κρίση, θα πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο στη διαβίωμαθηση και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων και πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ σκληρότερα προκειμένου να επιτύχουμε του στόχου που έχουμε θέσει. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο συζητάμε πολύ συχνά εδώ στην Επιτροπή και επηρεάζει το θέμα αυτό είναι η κινητικότητα της γνώσης. Ε, και ξέρετε ότι όλοι είμαστε υπέρ της κινητικότητας. Ε, θεωρούμε ότι μπορεί να ενισχύσει τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ένα καλύτερο μέλλον και μπορεί να οδηγήσει και στην καινοτομία και σε γενικές γραμμές ε, θεωρείται κάτι πάρα πολύ χρήσιμο, το οποίο έχει ε, πολύ σημαντικά ωφέλη και για τους ε, ανθρώπους μεμονωμένα, αλλά έχει ωφέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να προωθούμε την ε, κινητικότητα της γνώσης. Αυτό συμπεριλαμβάνεται και στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι μάλλον όλοι συμφωνούμε από αυτού. Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και νέες δεξιότητες και νέες θέσεις εργασίας. Η οικονομική κρίση ε, λογικά μείωσε την, ε, τη ζήτηση για κάποιες δεξιότητες ε, κάποιες τέτοιες τάσεις ήταν σαφείς πολύ πριν την οικονομική κρίση και μειώνεται συνεχώς ένα ποσοστό ανθρώπων που ζητάει νέες δεξιότητες. Η νέα τεχνολογία της γνώσης ζητά πολύ ψηλότερο σημείο εξειδίκευσης σε άλλα στοιχεία. Γι' αυτό λοιπόν Η υψηλή εξειδίκευση αυξάνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 29% στο 2008 στο 35% το 2010. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν πόσο πολύ χρειαζόμαστε υψηλού επίπεδου δεξιότητες. Ε, επίσης, προτείνονται κάποια στοιχεία στην ανακοίνωση και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι προκειμένου να επιτευθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει, υπάρχουν κάποιοι τρόποι να εργαστούμε προτείνουν για παράδειγμα το Συμβούλιο Παιδείας ε, να επικεντρωθεί στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και στο στόχο και τη στρατηγική του 2020 σε κάθε συνεδρίαση που θα κάνει. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στις συναντήσεις που θα γίνουν στο εξάμεινο το επερχόμενο. Το Συμβούλιο θα μπορούσε να εξετάσει το Μάρτιο παραδείγματος την κατάσταση και θα μπορούσε να διερευνήσει τα κοινά θέματα και να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα από τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης. Επομένως θα μπορούσε να υπάρχει ένα, ένα συνεχιζόμενο πρόγραμμα το οποίο θα οδηγεί και στην παρακολούθηση των, ε, θετικών, των εθνικών προγραμμάτων. Χρειάζεται επίσης να δούμε για με ποιο τρόπο θα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ώστε όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται να μπορούν να συνεργάζονται για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν προβλήματα πράγματι σε πολλά από αυτά τα θέματα που συνδέονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση και δεν έχουμε πάντα λογικές λύσεις και αυτό πρέπει να εξεταστεί. Υπάρχει και η αλληλοδιδακτική, όπως λέγανε παλιά, ή η διταχή μέσω ομοτήμων. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο η Δανική Προεδρία έχει δημιουργήσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου με στόχο να δημιουργήσει μια πολυεπίπεδη και πολυμερή προσέγγιση. Χρειάζεται λοιπόν να εργαστούμε σε περισσότερη λεπτομέρεια για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν αυτά στην πράξη. Αλλά υπάρχει μια πραγματική ανάγκη όλα τα προγράμματα αυτά και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η στρατηγική σκέψη να συνενωθούν κάπως και να εργαστούν καλύτερα και έχει τονιστεί ότι πρέπει να έχουμε μια καλύτερη σύνδεση μεταξύ της Ευρώπης 2020 και της εκπαιδευτικής Ευρώπης 2020 και πρέπει η Κομισιόν να οργανώνει κάθε χρόνο μια ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εμπλεκομένων στον τομέα της εκπαίδευσης και ε, κατά της και να δημιουργήσει ένα, προ, ένα φόρουμ για να εξετάσει την πρόοδο στην βελτίωση και τον εξυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατά της. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι μπορεί να γίνει ίσως πιο εύκολα από τα άλλα πράγματα τα οποία προτείνεται. Η Κομισιόν προτείνει επίσης να επικαιροποιεί τους δείκτες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης για να εξασφαλίσει ότι αυτοί που χρησιμοποιούνται για την καταμέτρηση της πρόοδου είναι συμβατοί με τους στόχους. Γι' αυτό η Κομισιόν θα παρουσιάσει ένα νέο σύστημα εποπτείας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ένα ελπίζουμε σύντομο έγγραφο για την δημιουργία ε, κυρίων δικτών και benchmarking για την ε, Ευρώπη του 2020 και τους στόχους Ναυαρχίδος για το 2020 στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να κινητοποιηθούν για να επιτύχουν τους στόχους οι οποίοι αναφέρονται στα προγράμματα της Ευρώπης 2020. Περιλαμβάνει λοιπόν την διαβίου εκπαίδευση, το πρόγραμμα Έρασμος για όλους και όλες, όπως θα είναι γνωστό στο μέλλον που πρέπει να συμπεριληφθεί εδώ και επίσης την χρήση των διαφορετικών πόρων για να εξασφαλίσουμε ότι όλες οι πτυχές της χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθούν και θα τεθούν στην καλύτερη δυνατή χρήση για να επιτευχθούν οι στόχοι εκπαίδευση και κατάρτιση στο φω ιδιαίτερος τη εκπαίδευση και τη κατάρτιση για να βγούμε από τη λούμπα τη τωρινή κρίση ή τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να βγούμε από την τωρινή κρίση. Αυτά λοιπόν όσο πιο σύντομα μπορούσα. Είναι αυτά που λέει η ανακοίνωση της Κομισιόν. Θα χρειαστεί να υπάρξει φυσικά πολλή συζήτηση για τα θέματα αυτά. Και αυτό είναι ένα πρωτόλιο επίπεδο ανταλλαγής απόψεων. Υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που έχουν ήδη λεχθεί. Μιλήσαμε για την ε, πρόορη σχολική εγκατάλειψη και το αναφέρει και η Κομισιόν και εμείς θα πρέπει να τονίσουμε και την ανάπτυξη της προσχολικής ηλικία, γιατί εδώ υπάρχει πολλή έρευνα όπως ξέρετε που δείχνει ότι αυτό που συμβαίνει στα παιδιά όταν είναι πολύ μικρά τα συνοδεύει σε όλη τη μεταγενέστερη ζωή τους και αν ξεκινήσουν με κάποιο χάντικαπ, αυτό το χάντικαπ δεν μπορούν να το ξεπεράσουν εύκολα, εξακολουθούν να έχουν απόδοση που δεν φτάνει την πραγματική τους δυναμικότητα και επειδή στο μέλλον η οικονομία θα βασίζεται όλο και περισσότερο στη γνώση. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να είναι κομμάτι τη έκθεση και να τύχει μεγαλύτερη έμφασης. Για τη διαβίου. Εκπαίδευση. Ε, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ότι σταματάει όταν κάποιο πάρει σύνταξη. Έτσι είναι η εντύπωση, αυτή είναι η εντύπωση που προκύπτει από αυτή την έκθεση, ότι κάποια στιγμή στα 64 τελειώνει η διαβίου μάθηση. Δεδομένου όμως ότι όλοι ζούμε περισσότερο και εργαζόμαστε και περισσότερο, δεν φαίνεται πολύ λογικό. Θα ήθελα να σκεφτούμε την παράταση της διαβίου μάθησης και για ανθρώπους ε, στη σύνταξη, που έχουν συνταξιδοτηθεί. Και κάτι άλλο, η εκμάθηση γλωσσών. Δεν είναι δυνατόν να πετύχουμε πολύ στην κινητικότητα αν ε, οι εργαζόμενοι μας, οι νέοι μας, οποιοδήποτε άλλους δεν έχει επαρκείς γλωσσικές γνώσεις και δεν μπορεί να επικοινωνήσει. Συνεπώς, δεν θα πρέπει απλώς να ενθαρρύνουμε, αλλά να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν ε, την διδασκαλία σύγχρονων ξένων γλωσσών. Έτσι ώστε η κινητικότητα να γίνει πραγματική πραγματικότητα, να γίνει ρεαλιστική η πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ιδιαίτερο πρόβλημα, ιδιαίτερα πρόβλημα στον Ηνωμένο αλλά είναι πρόβλημα και σε άλλα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να συνεχίσουμε να ε, υπογραμμίζουμε αυτή την έλλειψη. Αυτές είναι οι αρχικές μου σκέψεις ε, ως αντίδραση στην έκθεση της στην πρόταση της Κομισιόν. Πρέπει να προβάλλουμε καλύτερα ορισμένα πράγματα, τις ε, πολιτικές, ε, ε, την εφαρμογή, τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορεών και θεσμικών οργάνων, η εκπαίδευση και η κατάρτιση θα αποτελέσει κλειδί για την έξοδο από την οικονομική κρίση και εμείς έχουμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο σε αυτό. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Κύριος Κέλλη. Καταρχήν, ευχαριστώ την Μέρι Χόνιμπολ για, για αυτές τις παρατηρήσεις. Δεν θα μπορούσε κανείς να διαφωνήσει νομίζω με όσα είπε. Όλα όσα είπε είναι κέρια και θα βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020 αλλά και μετά. Ένα-δύο σχόλια θέλω να κάνω μόνο. Έχει δίκιο η μέρη που υπογραμμίζει τη σημασία της κατάρτισης. Το θέμα όμως είναι αν το πρόβλημα είναι όμως όταν οι διδάσκοντες δεν έχουν επαρκή προσόντα ή τα προσόντα τα οποία ε, μεταφέρουν και διδάσκουν δεν είναι τα κατάλληλα για τους καιρούς. Μέσω του, ε, παγκόσμιου προγράμματος, ε, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Παγκοσμιοποίησης στην Ιρλανδία ε, υποτίθεται θα διδασκόντουσαν καινούριε δεξιότητε, καινούρια πράγματα και στην πραγματικότητα μείναμε στα παλιά, στα παραδοσιακά. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θα πρέπει η κατάρτιση να συμβαδίζει με αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, με αυτά τα οποία θα χρειαστούμε στο μέλλον, τις δεξιότητες και τις ε, ε, ε, θα χρειαστούμε. 16 εκατομμύρια νέε θέσει εργασία θα δημιουργηθούν τα επόμενα χρόνια, όπω είπε, για ανθρώπους με νέες δεξιότητες, ενώ 12 εκατομμύρια θα χαθούν για ανθρώπους με παλαιές δεξιότητες. Συνεπώς είναι προ όφελο μας και απολύτω απαραίτητο να κάνουμε αυτή τη μετάβαση στις νέες δεξιότητες, στα νέα προσόντα. Επίσης, με την εξέλιξη τεχνολογίας, σχεδόν όλε οι νέε θέσει εργασία από εδώ και πέρα θα απαιτούν ε, διαρκή ενημέρωση και διαβίου Και αυτό θα πρέπει να το παρακολουθούμε ενδεχομένω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελευταίο μου σχόλιο. Η επαγγελματικός προσανατολισμός για νέους στα σχολεία. Αναρωτιέμαι, αυτοί που παρέχουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό στα σχολεία γνωρίζουν πού βρίσκονται οι ευκαιρίε άραγε, πού θα βρίσκονται στο μέλλον. Γνωρίζουν τι θα γίνει μέχρι το 2020 στους διάφορους κλάδους, επαγγελματικούς κλάδους. Μπορούν να πούνε στους νέους «Ε, σε, να, αντί να ακολουθήσουν μια παραδοσιακή πορεία να κάνουν κάτι άλλο. Μήπω το μόνο που κάνουν είναι να του λένε αφού έχει αρκετά καλή βαθμολογία για την νομική πήγαινε στη νομική ή για ιατρική πήγαινε στην ιατρική. Ξέρουμε για παράδειγμα εμεί ότι θα δημιουργηθούν 400.000 νέε θέσει ...στο στον τομέα τη ενέργεια. Αυτοί που παρέχουν επαγγελματικό προσανατολισμό το ξέρουν, το διδάσκουν, ε, κατευθύνουν του νέου προ τέτοιου είδου ευκαιρίε. Αυτό θα πρέπει να διασφαλίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και έτσι θα πετύχουμε. Ασφαλώς έτσι θα αυξήσουμε την απασχόληση, θα βελτιώσουμε το βιωτικό επίπεδο και θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί ε, ως Ευρώπη. Ευχαριστώ. Κανένα άλλο δεν θέλει να λάβει το λόγο. Θα ζητήσω από την Κομισιόν λοιπόν να λάβει το λόγο. Κύριε σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Τρούπελ. Θέλω να πω στην Κομισιόν και, και στην Συγήτρια ότι σας υποστηρίζουμε απόλυτα σε σχέση με την εκθεσία αυτή γιατί είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό μέσα στο χρονισμό της στρατηγικής 2020 να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Ήθιστε εδώ και δύο-τρία χρόνια να λέμε ότι ποτέ η παιδεία δεν ήταν τόσο ψηλά στη στρατηγική της Ευρώπης 2020. Νομίζω ότι είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αλλά θέλω να σας διαβιβάσω και το μήνυμα ότι δεν είναι κάτι που είναι μονάχα σε επίπεδο αρχών, αλλά και σε επίπεδο συγκεκριμένων και αυτών αποτελεσμάτων. 16 χώρες πέρυσι πήρανε ειδικέ αναχώρα συστάσεις που συνδέονται ούτως ή άλλως με την παιδεία και ενεκρίθησαν από τους αρχηγούς κυβερνήσεων και σε σχέση με τα οποία ήδη τον Απρίλιο πρέπει να κάνουν μια έκθεση για την πρόοδο που επιτύχαν. Αφορούν μερικέ φορέ την προορισχολική εκμετάλλευση, την, άλλες φορές την κατάρτιση, την επαγγελματική ή τη διαβίου, ε, εκπαίδευση, αλλά σε επίπεδο αρχηγών κρατών θεωρείται σημαντική η τη διαβιου εκπαιδευση αλλα σε επιπεδο αρχηγων κρατων θεωρειται σημαντικη η παιδεια ένα άλλο στοιχείο προέρχεται από την προηγούμενη συζήτηση για την κινητοποίηση των διαφθορτικών ταμείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παιδεία να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πόροι και για την κουλτούρα. Εδώ συζητάμε για την παιδεία. Οι προτάσεις που έχει κάνει η Κομισιόν για τους επόμενους διαρθρωτικούς πόρους, ιδίως το Κοινωνικό Ταμείο, ε, τονίζουν ιδιαίτερα το θέμα της παιδείας και το τρίτο θέμα ανέφερα προηγουμένως <clears throat> όταν ήθελα να βοηθήσω τον νέο μου συνάδελφο. Σε 8 χώρε που έχει μεγάλη ενεργεία στείλαμε ομάδε εμπειρογνωμόνων για να συζητήσουν με του υπουργού παιδεία και απασχόληση και του υπουργού οικονομικών βεβαίω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να ανακινητοποιήσουμε ορισμένα κονδύλια των ταμείων αυτών που δεν χρησιμοποιούνται, παραδείγματο χάρη στην Ισπανία αλλά και να δούμε πώς μπορούμε οι καλές πρακτικές ορισμένων χωρών να είναι χρήσιμες και σε άλλες χώρες. Παραδείγματος, και το ξέρετε ο κύριο Τρίπελ, το αυστριακό σύστημα, το διτό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης που ισχύει και στη Γερμανία και στην Δανία, που είναι απαραίτητο για την μετάβαση από τον, χώρο παιδεία στο χώρο εργασία πρέπει να σα πω ότι σε αυτές τις αποστολές η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία, οι χώρες που είναι πολύ ψηλή η ανεργία στις, στις αυτές τις χώρες, αποφασίστησαν να εμφορείται η εκπαιδευτική τους πολιτική από το διτό σύστημα της Αυστρίας, Γερμανίας και Δανίας. Αποφασίσαν να εμπνέονται από αυτό γιατί πρέπει να το προσαρμόσουν στη χώρα και την κουλτούρα. Αλλά αυτό είναι ακριβώς η συνεργασία μεταξύ των χωρών, όχι μόνο για να εκπονούμε έγγραφα, αλλά για να χρησιμοποιούμε τις βέλτιστες πρακτικές, να τις μεταλαμπαδεύουμε και να τις εφαρμόσουμε στις χώρες που είναι απαραίτητο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η Κομισιόν έκανε την έκθεσή της για την εφαρμογή αυτής της συνεργασίας που στρέφεται και προς το παρελθόν τα τρία τελευταία χρόνια, τι έγινε τότε και υπάρχουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες έλαβαν χώρα, ιδίως για τη σχολική εγκατάλειψη και εκεί το Συμβούλιο ενέκρινε μια σύσταση που είναι πολύ σημαντική, αλλά επίσης και μελλοντόστροφα στοιχεία. Γιατί απέχουμε πόρο και παρασάγκα του στόχου που δεν είναι και τόσο φιλόδοξος, δηλαδή 10% μοναχασχολικής εγκατάλειψης στην Ευρώπη, ενώ είμαστε στο 14%. Πρέπει λοιπόν οι εθνικές στρατηγικές να εφαρμοστούν καλύτερα. Επίσης, Αναφερθήκαμε στο επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου ο στόχος μας είναι πολύ φιλόδοξος, 40% των νέων να έχουν πανεπιστημιακά διπλώματα και πλησιάζουμε. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο να διατρέξουμε, ιδιαίτερα σε ορισμένε χώρες. Η κυρία η η κυρία Honeyball, αναφέρθηκε στην διαβίου εκπαίδευση. Την εκπαίδευση ενηλίκους δείχνουν οι δείκτες ότι υπάρχει λιγότερη εκπαίδευση των ενηλίκων από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Ενώ ο πληθυσμό γυράσκει, δεν γυράσκει διδασκόμενο. Ενώ πρέπει να εργάζεται περισσότερο, δεν υπάρχει περισσότερη διαβίω εκπαίδευση. <coughs> Εδώ οι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορούν να μα βοηθήσουν. Προτεραιότητε. Στρέφονται και προ το παρελθόν τα προηγούμενα τρία χρόνια, αλλά και το μέλλον τα δύο-τρία επόμενα χρόνια πρώτη προτεραιότητα μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην παιδεία. Επιμένω εδώ γιατί αυτό το οποίο γίνεται στα κράτη-μέλη και είναι καινούριο. Συζητάμε το θέμα της χρηματοδότησης της παιδείας. Όχι μόνο σε επίπεδο πανεπιστημίου, αλλά σε όλα τα επίπεδα. Λέμε ότι πρέπει εγκαίρως να υπάρξει επένδυση και να υπάρξει επένδυση στην αρχή της σχολικής εκπαίδευσης. Μιλήσατε για το early child care. Είναι πολύ σημαντικό και για τους πληθυσμούς των μεταναστών να μπορούν το ταχύτερο δυνατό να έχουν την πρόσβαση στην παιδεία αυτή. Υπάρχουν λοιπόν οι επενδύσεις για, τον, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να είναι στο κέντρο των συζητήσεων στα επόμενα 2-3 χρόνια και αν μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας βοηθήσει στον τομέα αυτό θα είναι καλό δεχτό. Δεύτερη προτεραιότητα, σχολική εγκατάλειψη. Και επίσης η επόμενη προτεραιότητα στη συζήτηση είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων, skills στα αγγλικά. Δεξιότητες που να προσαρτολίζονται καλύτερα προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σημαντικό με την ε, μεγάλη ενεργεία που έχουμε τώρα, αλλά και δεξιότητες οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κοινωνίας του 21ου αιώνα. Και αναφέρθηκαν ιδιαίτερα οι δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τις νέες τεχνολογίες ή δεξιότητες που θα οδηγήσουν σε μια δημιουργική και δημιουργούσα θέσεις απασχόλησης και καινοτόμα Ευρώπη. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θέλουμε να εργαστούμε σε αυτά. Και η τελική μου παρατήρηση είναι απλώς να ζητήσω μια βοήθεια από τη δική σας πλευρά για αυτό που λέμε ευκυβερνησία. Στο Συμβουλίο Υπουργών όλο και περισσότερο οι Υπουργοί ενδιαφέρονται για τα θέματα ευρωπαϊκού προσανατολισμού της εκπαίδευσης. Θεωρούν όμως πολλές φορές ότι η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι κάτι το οποίο δεν τους απασχολεί σε άμεσο επίπεδο τουλάχιστον στις χώρες τους. Αυτό δεν ισχύει όλα αυτά που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βοηθήσουν την εθνική πολιτική. Αν μπορείτε λοιπόν να μας βοηθήσετε να κινητοποιήσουμε καλύτερα <clears throat> τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων και τα εθνικά κοινοβούλια. Έχουμε προτείνει να γίνει ένα φόρουμ για τα θέματα αυτά και μπορεί να υπάρχει μια ευρύτερη συμμετοχή. Έχουμε προτείνει την ε, ε αξιολόγηση από ομοτήμους, το peer review. Η Ισπανία που έχει αυτό το υψηλό, πολύ υψηλό επίπεδο σχολικής εγκατάλειψης θα συμμετάσχει σε αυτή την αξιολόγηση από ομοτήμους, από χώρες που είναι καλύτεροι, καλύτερα τα ποσοστά αυτά για να δει πώς αντιμετωπίζουν αυτές οι χώρες την ε, σχολική εγκατάλειψη και φυσικά και η έκθεση εποπτείας που δεν θα είναι ένα χοντρό βιβλίο με πάρα πολλές στατιστικές αλλά θα είναι αντίθετα ένα έγγραφο που θα βασίζεται στους πιο σημαντικούς δείκτες και αυτό είναι αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μερές. Θέλετε να πείτε κύριε Χάνεμπολ. Πολύ γρήγορα συντομία. Σύμφωνο απόλυτα με όσα είπε ο κύριο Σκέλη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε εγρήγορση για να καταρτίζουμε και τους καταρτίζοντες ε, έτσι ώστε και οι καταρτίζοντες να καταρτίζουν σωστά αυτούς που καταρτίζονται. Γιατί θα πρέπει οι νέοι να μαθαίνουν αυτά που χρειάζονται. Και οι καταρτίζοντες, οι διδάσκοντες ε, κάποια στιγμή έμαθαν ορισμένα πράγματα τα οποία θα πρέπει όμως να επικαιροποιούν. Οπότε ο κ. Σκέλη έχει πολύ δίκιο. Ευχαριστώ την Κομισιόν για όλες τις παρατηρήσεις. Δεν χρειάζεται να τις ε, σχολιάσω. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση προς το Κοινοβούλιο να λάβει μέρος στο φόρουμ που θα οργανώσει η Κομισιόν και στην διαδικασία αξιολόγησης από ομοτήμους αν χρειάζεται η συμμετοχή μας εκεί. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστούμε για όλα αυτά και να βρισκόμαστε σε συνεχή διάλογο. Γιατί τελικά ο στόχος είναι κοινό. Και σε άλλα, και σε άλλα συνέδρια αν μας καλέσετε θα έρθουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάνιμπολ. Θα έχουμε την παρουσίασή σας της, ε, του σχεδίου έκθεσης τον Απρίλιο. Σημείο 16 η έγκριση των ε, αποφάσεων των συντονιστών. Συναντήκα σήμερα το πρωί και οι αποφάσεις σας έχουν σταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Και η επόμενη συνεδρίαση. Μπορείτε να εγκρίνετε καταρχήν τα... Ωραία, εγκρίνετε τα συμπερασματών των συντονιστών. Σημείο 17. Υπάρχει κάτι άλλο, ένα άλλο θέμα που θέλετε να γίνετε. όχι. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συμμετοχή σας και ιδίως τους ε, μεταφραστές μας και η επόμενη συνεδρίασή μας είναι 27 Μαρτίου. Καλό βράδυ. So,